ο πρόεδρος Βόμποντα δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και με όρισα να προεδρεύσω αλλά αυτό δεν θα είναι δύσκολο γιατί η ποιότητα των συμμετεχόντων και της γραμματείας είναι δεδομένη. Ευχαριστώ να κάνετε ησυχία στο βάθος και να διευκολύνεται τις εργασίες των διερμηνέων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν δύο σημεία, με δύο σημεία πρώτα, μιας και ε, δεν είναι εδώ ο κύριος Βόμποντα. Θα αναβάλουμε το 7 και το 12. Έχετε κάποιες αντιρρήσεις, όχι. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές και δεν υπάρχουν αγκυρίσεις. Ε, για την ημερήσια διάταξη, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνω τις εξής ανακοινώσεις. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Σας ακούω από τα ακουστικά μου. Έχετε ωραία φωνή, αλλά να μην σας ακούμε παρακαλώ. Στα διάφορα προτείνω να δώσουμε το λόγο στη νομική υπηρεσία, τον κύριο Κάιολα, να μας παρουσιάσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Μαΐου 14 για το c 658 Παύλα 1 για την διακρατική εταιρική συμφωνία με τον Μαυρίκιο. Αν δεν έχετε κάποιες αντιρρήσεις μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στα κανονικά σημεία της ημερήσιας διάταξης. Παρουσίαση λοιπόν της νομικής υπηρεσίας του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας και για τη νομική βάση και για τις ε, διαφορές της δικαστικές τις οποίες εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Ντρέσλερ, προϊστάμενος ε, της νομικής υπηρεσίας. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή σας για την πρόσκληση την οποία μας απίφθηνε που μας δίνει την δυνατότητα στην αρχή αυτής της νομοθετικής εντολής την δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της νομικής υπερουσίας και του υπηρεσία και του τρόπου που λειτουργεί. Εδώ έχω και την κυρία Μαρία Χωσέ Μαρτίνες Ιγκλέσιας που είναι διευθύντρια της νομικής υπηρεσίας, υπεύθυνη για νομοθετικά θέματα. Γνωρίζει πολύ καλά την Επιτροπή αυτή, γιατί εργάστηκε στη γραμματεία σας για πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω συγγνώμη ε, εκ μέρους του άλλου διευθυντή, του Ρικάρντο Πάσος, που είναι υπεύθυνος για κοινοβουλευτικά και θεσμικά θέματα. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα ανάμεσά μας. Ε, ξεκινώντας λοιπόν κάποιους, ε, κάποια στατιστικά στοιχεία είναι γενική διεύθυνση, 111 οργανικές θέσεις, 70 ε, δικηγόροι και 41 ε, βοηθοί δικηγόροι. Γεωγραφικά είμαστε κομμένοι στα δύο. Το ένα τμήμα είναι στο Λουξεμβούργο και το άλλο τμήμα το οποίο ασχολείται με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, εδώ στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν τρεις διευθύνσεις. Η πρώτη, όπως είπα, είναι η διεύθυνση του Πάσος, θεσμικά και κοινοβουλευτικά θέματα. Η δεύτερη, της Μαρία Χωσέ, ε, και οι δύο καλύπτουν το σύνολο των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η τρίτη διεύθυνση έχει έδρα κυρίως στο Λουξεμβούργο και ασχολείται με διοικητικά, διαχειριστικά και οικονομικά θέματα. δηλαδή θέματα υπηρεσιακού κανονισμού, ε, συμβάσεις οικονομικές, κτίρια κτλ. Οι 28 εθνικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εκπροσωπούνται. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις γλώσσες και όλα τα νομικά συστήματα και τους νομικούς πολιτισμούς των κρατών μελών στην υπηρεσία μας. Η νομική υπηρεσία ως έχει δημιουργήθηκε το 1986 επισήμως, γιατί φάνηκε απαραίτητο στη δεδομένη φάση να υπάρξει μία λοιπόν νομική υπηρεσία, διότι υπήρχαν όλο και περισσότερες ε, νομικές αρμοδιότητες, οι οποίες ε, δημιουργήθηκαν προοδευτικά από τις αλλαγές της συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπογράμισε το καθήκον που έχουν τα θεσμικά όργανα να αντιμετωπίζουν τις, τη διαχείριση των υπηρεσιών τους και στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης νομικής υπηρεσίας η οποία να δίδει συστάσεις και συμβουλές ανεξάρτητες και δίκαιες. Σχετικά με τη δική μας υπηρεσία υπάρχει πάντα ένας δικηγόρος της νομικής υπηρεσίας που παρακολουθεί τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχουμε τον Ντάνιελ Βερά, ο οποίος είναι στο πίσω μέρος της αίθουσας, και την κυρία Πάνσεβα, η οποία παρακολουθεί τις δραστηριότητες της δικής σας επιτροπής. Είναι αυτονόητο ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, δεδομένων των αρμοδιοτήτων της, έχει ειδικέ νομικές αρμοδιότητες. Παράλληλα με τις αρμοδιότητες αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημο 6, καλύπτουμε εταιρικό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα, αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, ε, συνεργασία δικαστικού και ε, διοικητικού ε, και θέματα που άπτονται των και κάποιων άλλων αρμοδιοτήτων ε, για το όργανο αυτό. Ανάμεσα σε αυτές τις αρμοδιότητες υπάρχει ο έλεγχος της επικουρικότητας, της αναλογικότητας στα θέματα των νομικών βάσεων και εδώ η Μαρία Χωσέ θα καλύψει το θέμα το έχετε και στην ημερήσια διάταξή σας σήμερα, τον κατεξουσιοδότηση πράξεων, των εφαρμοστικών πράξεων, της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας, της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και τέλος, την προστασία των δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι αρμοδιότητες αυτές λοιπόν αποτελούν ένα σημαντικό ρόλο για την υπηρεσία μας και συνεισφέρουν στον σεβασμό της αρχής της νομιμότητας και κράτους δικαίου. Σε αυτό άλλωστε και το πλαίσιο θα ήθελα να αναφερθώ τώρα για τις διαφορετικές αποστολές της νομικής υπηρεσίας. Η νομική υπηρεσία έχει ένα διτό θα έλεγα ρόλο πρώτον είναι ο παροχέας νομικών συμβουλών προς το κοινοβουλευτικό όργανο. Δεύτερον, υπερασπίζεται το όργανο αυτό σε δικαστικό επίπεδο. Αυτός είναι ο ρόλος της νομικής υπηρεσίας. Τώρα για την πλευρά των συμβουλών και συστάσεων είναι οι συγκεκριμένοι δικηγόροι που εργάζονται σε μας και οι οποίοι παρακολουθούν τις εργασίες των πολιτικών σώματων και δίδουν ημερήσιες ανεπίσημες συμβουλές και συστάσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, στην γραμματεία και, στα κρατη και στους βουλευτές συγγνώμη, μεμονωμένα, ιδιαίτερα όταν είναι ε, εισηγητές ή σκιώδεις εισηγητές σε θέματα νομοθετικά. Πολλές φορές όμως οι ερωτήσεις έχουν πολλαπλό χαρακτήρα, δύσκολο και σύνθετο και δεν μπορεί να απαντηθούν από μια ανεπίσημη πηγή. Ως εκ τούτου εκεί μπορεί να απαιτηθεί μια επίσημη νομική σύσταση. Η σύσταση αυτή μπορεί να ζητηθεί από τα κοινοβουλευτικά σώματα, τον Πρόεδρο, το Προεδρείο, την διάσκεψη των Προέδρων, τους α, ε, κοσμήτορες και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Μπορεί να ζητηθεί γύρω από τη θέμα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Όταν έχετε ένα θέμα δηλαδή για το οποίο θα θέλατε να υπάρξει μια επίσημη νομική σύσταση ή συμβουλή, μπορεί να ζητηθεί μέσω του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Οι συστάσεις τις οποίες παρέχει η νομική υπηρεσία ε, έχουν σαν στόχο ε, να διευκολύνονται οι νομοθετικές δραστηριότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο δεύτερος ρόλος τώρα της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων αφορά την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δικαστικό επίπεδο και θα συνεχίσω στην γαλλική γλώσσα πλέον και όχι την αγγλική. Όταν υπάρχουν δικαστικές διαφορές σαν όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και περισσότερο εμπλέκεται σε διαφορές οι οποίες συζητώνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, και σε εθνικά δικαστήρια. Il existe différents cas de figure, mais le rôle de la commission juridique est toujours ο ρόλος της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ε, σημαντικός. Σε ένα πρώτο σενάριο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατηγορούμενο. Σε αυτή την περίπτωση σύρεται στα πλαίσια μιας νομικής δικαιοδοσίας. Πρόκειται πολλές φορές για μια ακύρωση μιας πράξης την οποία έχει ψηφίσει ή ε, αμφισβητείται ο σεβασμός των συμβατικών ή και εξωσυμβατικών υποχρεώσεων του. Σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο δεν έχει επιλογή, πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό του και ζητά από την νομική υπηρεσία να το κάνει. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή όταν ακριβώς το Κοινοβούλιο θέλει να ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία, τότε ο ρόλος της νομικής επιτροπής του Κοινοβουλίου είναι κυρίαρχος. Αυτό περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου στο άρθρο 141. Για να συνδράμει λοιπόν τη νομική επιτροπή, η νομική υπηρεσία παρέχει πάντα μια ανάλυση της υπόθεσης περί γίνεται η ε, συζήτηση. Ε, στην πρώτη περίπτωση λοιπόν όταν το κοινοβούλιο προσφεύγει στα δικαστήρια έχει την δυνατότητα να ζητήσει μια προσφυγή επί παραλήψη εις βάρος πράξεων άλλων θεσμικών οργάνων οι οποίες θα έχουν συνέπειες νομικής φύσεως εις βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, στην ουσία όταν αμφισβητούνται τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν υπάρχει πολλές φορές πρόβλημα νομικής βάσεως και εδώ η συνάδελφος ε, Μαρτίνες θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό μπορεί να συμβεί επίσης όταν υπάρχει παραβίαση των αρμοδιοτήτων, των κανόνων που διέπουν τις αρμοδιότητες όταν υπάρχει η παραβίαση μιας βασικής αρχής ενός θεμελιώδους δικαιώματος ε, σαν παράδειγμα της αρχής της επικουρικότητας κτλ. Όταν υπάρχει μια παραβίαση του κοινοτικού δικαίου που απαιτεί από το Κοινοβούλιο να ζητήσει την ακύρωση της νομικής πράξεως, ε, τότε ο πρόεδρος θα πρέπει να ζητήσει από τη νομική υπηρεσία να κάνει ε, τις κατάλληλες ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επλακεί και η Ολομέλεια εφόσον ο πρόεδρος δεν ακολουθήσει τη σύσταση της Επιτροπής σας. Μια άλλη περίπτωση, όταν πρόκειται να κατατεθούν παρατηρήσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Πρόκειται για θέματα τα οποία έχουν, ε, εκπροσωπούνται διαφορετικά συμφέροντα, υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο διαφορετικές ερμηνείες μια εθνική δικαιοδοσία θέτει θέμα ερμηνείας και εγκυρότητας μιας πράξης την οποία αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή συναποφάσισε πολύ συχνά. Σε αυτή την περίπτωση η νομική ε, επιτροπή νομικών υποθέσεων ε, προτείνει την παραπομπή του θέματος στα δικαστήρια έτσι ώστε να υπάρξει η συζήτηση στο συγκεκριμένο επίπεδο, ιδιαίτερα όταν αμφισβητείται η εγκυρότητα η νομική μιας αποφάσεως του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης και τη δυνατότητα παρέμβασης σε διαφορές τις οποίες δεν είναι το κύριο μέρος. Μπορεί να υπερασπιστεί σαν παράδειγμα να συνδράμει είτε αυτόν ο οποίος προσφεύγει είτε αυτόν ο οποίος κατηγορείται κάθε φορά. Αυτό μπορεί να αφορά την νομιμότητα μιας πράξης στην επεξεργασία της οποίας πήρε μέρος το Ευρωπαϊκό να απειλούνται οι αρμοδιότητές του. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σε στενή επικοινωνία με την γραμματεία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ε, σεβόμενη και τις ε, προθεσμίες, της χρονικές, οι οποίες ε, είναι μερικές φορές ιδιαίτερως δεσμευτικές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείται από συγκεκριμένους ε, υπαλλήλου οι οποίοι ορίζονται από τον Juris Consultus μετά από οδηγίες του Προέδρου. Ε, αυτοί γνωρίζουν τις διαδικασίες, σέβονται τις διαδικασίες και παρουσιάζουν τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει μονίμως ε, σταθερά θεσμικό χαρακτήρα διότι εκπροσωπεί το σύνολο του οργάνου μας. Η υπεράσπιση είναι νομικής φύσεως με αποκλειστικά νομικά κριτήρια και, με, και όχι με πολιτικές σκέψεις και αιτιολογίες. Ε, όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια των κανόνων που αποφασίζει το Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο και αυτό αφορά το σύνολο των δικηγόρων που μετέχουν στις διαδικασίες του. Συμπερασματικά, για να μην σας καθυστερήσω πολύ, να θυμίσω ότι οι στόχοι της νομικής υπηρεσίας είναι διτής φύσεως. Πρώτον, προάσπιση των συμφερόντων του οργάνου και δεύτερον, να προσφέρουμε στα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία νομική συνδρομή υψηλής ποιότητας Γι' αυτό λοιπόν και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που τρέφετε στην ε, γραμματεία μας, όπως επίσης και να ευχαριστήσω τη γραμματεία σας για την εξαιρετική μορφή συνεργασίας την οποία μας παρέχει. Είμαι στη διάθεσή σας και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρτίνες Ιγλέσιας για να μας παρουσιάσει το θέμα των νομικών βάσεων για πέντε λεπτά παρακαλώ. Θα προσπαθήσω, λέει η κυρία Ιγλέσιας. Οι δικηγόροι είναι συνοπτικοί, αν στην έκφρασή της. Όπως λοιπόν το είπε και ο Γιούρις Κονσούλτους, το κανονισμός του Κιβουλίου παρέχει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εγκάρσιες αρμοδιότητες των οποίων βασικός στόχος είναι να δοθούν εγγυήσεις για την ποιότητα της νομοθετικής δραστηριότητας και τη διασφάλιση της νομικής βεβαιότητας. Όταν προβλέπεται η λήψη μιας πράξης νομικής, θα πρέπει να είμαστε καταρχάς βέβαιοι ότι έχουμε τις αρμοδιότητες που απαιτούνται και τις εξουσίες για να το κάνουμε. Δεν έχουμε πλήρεις αρμοδιότητες και εξουσίες. Ε, η συνθήκη είναι αυτή η οποία ορίζει κάθε τομέα αρμοδιότητας. Αυτό αναγνωρίζουμε λοιπόν σαν βασική αρχή κατανομής αρμοδιοτήτων. Οι ρήτρε της συνθήκης που δίδουν στην Ένωση τις εξουσίες είναι οι λεγόμενες νομικές βάσης. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της συνθήκης το εκφράζουν αυτό λέγοντας ότι το εύρος και ο τρόπος εφαρμογής των κοινοτικών αρμοδιοτήτων καθορίζονται από τις προβλέψεις της συνθήκης τις σχετικές με κάθε τομέα. Δηλαδή δεν αρκεί ένα θέμα να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει το άρθρο 3 έτσι ώστε το θέμα αυτό να περιληφθεί αυτόματα στους στόχους που εκφράζει η συνθήκη ή έτσι ώστε να μπορεί ε, άκρητα να παίρνει αποφάσεις ο νομοθέτης είναι απαραίτητο ένα συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης να το ορίζει αυτό, να το επιτρέπει αυτό και ως προς τη διαδικασία και ως προς τους τρόπους δράσης της Ένωσης. Αυτά όλα είναι αυτό που λέμε η νομική βάση. Ε, δεν εκπλήσεται λοιπόν κανείς όταν βλέπει ότι το Κοινοβούλιο προβλέπει ένα δίκτυο ασφαλείας το οποίο συγκεκριμενοποιείται από την έλεγχο και την επαλήθευση που κάνει σε επίπεδο νομικής βάσης η νομική υπηρεσία. Κάθε τροποποίηση της νομικής βάσης όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί μία ε, προτεραιότητα γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής σας, ακόμα και αν η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι δεσμευτική. Παρ' όλα αυτά το Κοινοβούλιο κυρίαρχα η Ολομέλεια θα αποφασίσει, αλλά θα γνωρίζει περί ποιου αποφασίζει, γιατί υπάρχει πάντα μία σύνθεση των θέσεων της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων σε σχέση με τη νομική βάση. Γιατί δίνουμε τέτοιο βάρος στην εξέταση της νομικής βάσης. Το πρώτο είναι να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες δράσης σε συγκεκριμένους τομείς. Οι νομικές βάσεις αυτές καθορίζουν και άλλα χαρακτηριστικά της κοινοτική δράσης. Το Κοινοβούλιο, το τι θα κάνει πρώτον και με ποιες διαδικασίες. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε τομείς διαδικαστικούς γιατί καθορίζονται οι ε, δικές τους αρμοδιότητες. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι στο παρελθόν όταν η συναπόφαση δεν ήταν ε, η κανονική συνήθις διαδικασία. Ε, πολλές φορές έτσι κι αλλιώς οι απλές επιλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν καθόριζαν από μόνες τους τη νομική βάση. Σύμφωνα με την ομολογία τη σταθερή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η επιλογή της νομικής βάσης θα πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες μεταξύ των οποίων ο στόχος και το περιεχόμενο της προτινόμενης νομικής πράξης. Αυτές τις φράσεις θα τις ακούσετε πάρα πολλές φορές όταν συζητάμε για τις νομικές βάσεις. Τώρα για τη διαδικασία. Το δικαστήριο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η διαδικασία από μόνη της δεν είναι ένα επιχείρημα έγκυρο. Είναι η συνέπεια των επιλογών που έχουν γίνει σε σχέση με τις αποφάσεις της πολιτικές που λαμβάνει σαν κοινοβούλιο. Ένα από τα πιο προβληματικά θέματα σε σχέση με τις νομικές βάσεις είναι όταν υπάρχουν ε, δύο ή περισσότεροι στόχοι και υπάρχουν δύο ή περισσότερες συνιστώσεις στο περιεχόμενό του. Εδώ το δικαστήριο μας δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Όταν υπάρχει ένα τμήμα του περιεχομένου το οποίο θεωρείται πιο σημαντικό και το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύριο, τότε η νομική βάση που του αντιστοιχεί είναι η νομική βάση της πράξης. Και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία σε έκτακτες περιπτώσεις όπου οι στόχοι των συνιστοσών ε, ε, μεταξύ τους είναι αλληλένδετες, τότε μπορεί να υπάρχει μια διπλή νομική βάση. Αυτό είναι όμως πολύ περίπλοκο απαιτείται οι δύο νομικές φάσεις να είναι συμβατές μεταξύ τους, να μην προβλέπουν διαδικασίες οι οποίες να είναι ασύμβατες, ασυνδίαστες. Η μία να θέλει την ομοφωνία με απλή ε, πλειοψηφία και η άλλη την συναπόφαση με ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Αν και μερικές φορές το δικαστήριο έχει αλλάξει ε, τις αποφάσεις αυτές. Λοιπόν συμπερασματικά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και παρέμβαση της υπηρεσίας μας σε σχέση με τη διπλή ή τριπλή νομική βάση. Αυτό καθορίζει έτσι και αλλιώς και τα μέσα. Κάποιες νομικές βάσεις επιτρέπουν κανονισμούς, κάποιες άλλες οδηγίες, κάποιες άλλες διαφορετικές νομικές πράξεις. Εφαρμόζοντας πάντα την αρχή της αναλογικότητας η οποία καθορίζει και την ένταση της κοινοτική δράσης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που καθορίζεται από τη νομική βάση είναι οι διαδικασίες της κοινοτική δράσης. Στον τομέα του περιβάλλοντος, σαν παράδειγμα, στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, πάρα πολύ συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει επιλογές. Στον τομέα του περιβάλλοντος τα κράτη-μέλη δεν έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν μάλλον αντίθετα, τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν πιο περιοριστικά μέτρα από αυτά τα οποία προβλέπει η κοινοτική απόφαση. Ενώ το ίδιο δεν ισχύει στην εσωτερική αγορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μερικές φορές κάποιες ε, δυσκολίες. Σήμερα το απόγευμα θα κληθείτε άλλωστε να πάρετε και μία απόφαση για μία νομική βάση, τη νομική βάση της σύμβασης ε, της, ε, για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Σύμβαση για τα απειλούμενα είδη πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται. Εδώ υπάρχουν δύο καταρχήν προτινόμενες νομικές βάσεις. Το Συμβούλιο ακύρωσε τη μία. Η Επιτροπή πρότεινε το εμπόριο και το περιβάλλον. Το Συμβούλιο ακύρωσε το εμπόριο. Θα κληθείτε λοιπόν να αποφασίσετε αν η επιλογή του Συμβουλίου είναι η κατάλληλη ή θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαφορετική διαδικασία. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη, στη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης. Όμως έχουν διαφορετική εμβέλεια. Το περιβάλλον είναι μια διαμοιραζόμενη αρμοδιότητα, μια κοινή αρμοδιότητα, ενώ το εμπόριο είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα της ε, Ένωσης και η συνθήκη εννοεί ότι οι απόλυτες αρμοδιότητες της κοινότητας δεν επιτρέπουν καμία δυνατότητα δράσης στα κράτη-μέλη. Και αυτό εξηγεί την επιλογή την οποία έκανε το Συμβούλιο. Ακύρωσε τη νομική βάση για το εμπόριο ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Συνεπώς, σας έδωσα το παράδειγμα για να σας δείξω τη σημασία που έχουν αυτά τα οποία αποφασίζεται. Πάντα η φύση, η βάση μάλλον μιας νομικής βάσης δεν είναι ε, παρά ένα άρθρο της συνθήκης, όχι το προερχόμενο δίκαιο, το δευτερεύον δίκαιο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα και για να σεβαστώ τις επιθυμίες του Προέδρου μας θα σταματήσω εδώ να σημειώσω ότι στα πλαίσια της ανάλυσης των νομικών βάσεων η νομική υπηρεσία σας είναι πάντα στη διάθεσή σας. Αλλά την απόφαση πάντα λαμβάνει το πολιτικό όργανο, η Επιτροπή δηλαδή, και η ευθύνη είναι δική σας. Και εμείς εδώ είμαστε για να διευκολύνουμε στο μέγιστο δυνατό τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι μια καταπληκτική, εντυπωσιακή βελτίωση των γαλλικών σας τα τελευταία χρόνια. Αυτό το παρατηρώ καλύτερα και από τα αγγλικά και από τα ισπανικά. Ε, έχει κανείς ερώτηση ή παρατήρηση σχόλιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο διαφορετικές κάπως ερωτήσεις έχω να θέσω γίνεται μεγάλη συζήτηση για καλύτερη ρύθμιση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η βάση για μια υγιή νομοθεσία, μια ε, ισότιμη αντιμετώπιση των θεμάτων και ήθελα να ρωτήσω τι θα συνέβαινε εάν υπήρχαν μέτρα εφαρμοστέα τα οποία θα έπρεπε να αναλάβουν την ε, ένταξη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση, τότε τι θα έκανε το Κοινοβούλιο μέσω της Νομικής Επιτροπής, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για να υπερασπιστεί αυτήν την νομοθεσία. Εάν δεν υπήρχε κάποια στήριξη η οποία δεν μπορούσε να ακολουθηθεί ε, βάσει του κανονισμού. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο φορά τη νομική βάση. Συμβαίνει ποτέ μήπως ένα νομικό εργαλείο να βασίζεται σε μια συγκεκριμένη νομική βάση και να εξελιχθούν τα πράγματα με τέτοιον τρόπο μέσα στο χρόνο ε, που να υπάρξει μια διπλή ή τριπλή νομική βάση όταν εξεταστεί το θέμα και έχω ένα παράδειγμα με τον κανονισμό ε, Timber ο οποίος αφορά την έκθεση Τίμπερ από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωπαϊκές χώρες που έχει ε, μία σχέση με την ε, με τον ένα χώρο lobbying για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πελατειακή σχέση που έχει με τους εκτός Ένωσης. Υπήρχε λοιπόν μια νομική βάση για αυτό το θέμα που βασιζόταν μια νομική βάση σε περιβαλλοντικά θέματα. Τώρα όμως χαράχτηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπορική πολιτική και γι' αυτό ρωτώ τι γίνεται όταν εξελιχθεί, όταν μπορεί να εξελιχθεί η νομική βάση. Θέλετε να απαντήσετε αγαπητοί συνάδελφοι. Ίσως μπορείτε να δείτε στο τέλος το σύνολο των ερωτήσεων, τις απαντήσετε όλες μαζί πώς θέλετε, κύριε Κουτέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ θετική παρουσίαση γιατί έχετε, ξέρετε πάρα πολλά πράγματα, εγώ είμαι σχετικά καινούργια εδώ. Είπατε λοιπόν κυρία μου ότι μιλήσατε για το γιατί το Συμβούλιο θέλει να διαγράψει ορισμένα θέματα και πρέπει να το πράξει. Ποιες θα μπορούσε να είναι οι επιπτώσεις πάνω σε αυτό. Ένα θέμα εφαρμογής, ένα νομικό πρόβλημα θα μπορούσε να, είναι, να προκύψει εάν δεν συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δύο νομικές βάσεις Δηλαδή ποια θα είναι η διαφορά αν υπάρχει μία νομική βάση ή δύο νομικές βάσεις. Τι επιπτώσεις έχει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτό το τελευταίο θέμα θα τις πάρω με διαφορετική σειρά τις απαντήσεις. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το τελευταίο θέμα το Κοινοβούλιο ε, από αυτού ε, ζητείται να δώσει τη συγκατάθεσή του. Τι σημαίνει αυτό, ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, πει ότι δεν συμφωνεί με τη νομική βάση του Συμβουλίου γιατί υπάρχει μία ας πούμε η περιβαλλοντική για το Συμβούλιο και μπορεί να πει ότι προτιμάει τις δύο νομικές βάσεις. Έχει αυτή τη δυνατότητα και μετά έχει την επιλογή να είναι υπέρ του να δώσει συγκατάθεση ή όχι εάν α, εγκρίνει την θέση αυτή, αν δώσει τη συγκατάθεσή του, τότε η συμφωνία μπορεί να εγκριθεί ακόμα και αν δεν αλλάξει η νομική βάση. Η μόνη δυνατότητα για το Κοινοβούλιο είναι να επιμείνει στην περίπτωση της νομικής βάσης. Η μόνη δυνατότητα αν θέλει δύο νομικές βάσεις είναι να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του. δεν παίρνω θέση ούτε για τη μία περίπτωση ούτε για την άλλη, αλλά οπωσδήποτε και στις δύο περιπτώσεις το Κοινοβούλιο μπορεί να αμφισβητήσει, να παραπέψει το θέμα στο δικαστήριο μετά το θέμα της νομικής βάσης. Σε ό,τι αφορά την στήριξη των επιπτώσεων νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει εγγραφεί στις συνθήκες. Στη συνθήκη υπάρχουν μια, υπάρχει μια πρόβλεψη η οποία λέει ότι θα πρέπει να στηριχτεί η δράση της ε, Ένωσης και μπορεί να υπάρχει ένα εργαλείο για να μπορέσει να στηρίξει αυτό, αυτό το, αυτά τα κίνητρα. Και οπότε αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να δικαιολογήσει αυτά τα κίνητρα, ίσως θα είναι απαραίτητο να δώσει αυτή την στήριξη ε, και πιστεύω ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο γιατί υπάρχει σχετική νομοθεσία, υπάρχει ένας κανονισμός να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ένα θέμα, να έχει αλλάξει το περιεχόμενο, να ζητάει εξήγηση και στήριξη των κινήτρων και τότε μπορεί να αρκέσει η νομική βάση η οποία πρέπει να εγκριθεί. Άλλοι, άλλες παρεμβάσεις έχετε πάρει όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως θα έπρεπε, είστε ικανοποιημένοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς ε, ε, κύριε ε, de Κύριε Νομικέ Σύμβουλε και εσάς κυρία μου για όλες τις ε, σύμβουλες που μας δώσατε και την ακρίβεια των λόγων σας κυρίως. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η παρουσία ε, του ε, κυρίου Άντωνη τη ΔΕΛ, Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Παρακαλώ καθίστε. Να σας βλέπουμε θέλουμε. Έχουμε ομιλία. Vous avez la parole. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να παρουσιάσω την εργασία των υπηρεσιών μας της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι παρόν σήμερα ο Γενικός, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας και εγώ τον αντικαθιστώ. Όπως ξέρετε ορισμένοι από σας. Υπάρχει αυτή η νέα γενική ε, διεύθυνση ε, κοινοβουλευτών υπηρεσιών της έρευνας ένα χρόνο πριν, πάνω από ένα χρόνο πριν και άρχισε να υπάρχει αυτή η υπηρεσία τον Νοέμβριο του 2013 και υπήρχαν μια σειρά από τέτοιες υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, στήριξης υπηρεσίες και κατά κάποιον τρόπο ενισχύουμε ορισμένους τομείς όπως τον τομέα της έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης για την έρευνα. Έχουμε... Ε, πολλά ε, μέλη που ταξιδεύουν, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους που ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μια υπηρεσία παροχής στοιχείων, ε, βιβλιοθήκες, πληροφόρηση κτλ. Τέτοιου είδους υπηρεσίες δίνουν ένα φάσμα, δίνουν ένα φάσμα δημοσιεύσεων ε, που είναι η δουλειά της υπηρεσίας έρευνας, όποια είναι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποια και να είναι την καλύπτουμε στην υπηρεσία έρευνας. Δίνουμε λοιπόν, παρέχουμε υπηρεσίες στα μέλη μας ε, και υπάρχει μια παλιά βιβλιοθήκη που ανήκει στην δεύτερη διεύθυνση. Αυτή η παλιά βιβλιοθήκη έχει αρχεία με διάφορες αιτήσει των πολιτών που τώρα έχουν όλες ε, καταγραφεί στα αρχεία και έχουν πάρει ε, αριθμούς στα αρχεία και το τρίτο μέρος της γενικής διεύθυνσης αυτής είναι μια διεύθυνση που υπήρχε και προηγουμένως δύο χρόνια πριν και που είχε σχέση με την στήριξη ε, των, επιπτώσεων και ε, είναι ο τρίτος πυλώνας, είναι ό,τι έχει σχέση με τον τρίτο πυλώνα ε, της, με αυτόν ασχολείται η Γενική Διεύθυνση στο τρίτο της μέλος. Λοιπόν. η, διεύθυνση αυτή είναι, που αφορά τις επιπτώσεις είναι μία από τις μεγαλύτερες και ξεκίνησε με διαφορετικούς τρόπους. Καταρχήν έχει αρχεία ε, για τους που προέρχονται από την νομική υπόθεση και από όλες τις υποθέσεις που πέρασαν από την ε, υπηρεσία νομικών υποθέσεων πριν από μερικά χρόνια ε, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει ένα ανεξάρτητο σώμα το οποίο να κάνει την αξιολόγηση των, ε, σε θεσμική βάση των κρίσεων της Επιτροπής και μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τη βοήθεια των αρμόδιων Υπουργείων δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η υπηρεσία για να στηρίζει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πέρα από αυτό γίνεται μια επιθεώρηση για το πώς ε, δουλεύει αυτά τα θέματα η Επιτροπή, ε, να ταυτιστούν όλες οι αδυναμίες ε, σχετικά με τις εργασίες, πώς υποβλήθηκαν όλες οι σχετικές προτάσεις και πώς διευκαιρεώθηκαν και για όλα αυτά χρειάζεται μια νέα νομοθεσία για να μπορέσει σύμφωνα με το άρθρο 225 της συνθήκες να ε, καλύψει όλα αυτά τα θέματα. Ε, που είναι μια ενημέρωση αυτό το άρθρο του παλιότερου σχετικού άρθρου της συνθήκης. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε στήριξη για τις επιπτώσεις και από την άλλη είναι παροχή ε, ερευνών για την υπηρεσία έρευνας. Όλα αυτά υπάρχουν εδώ και δύο χρόνια ή μάλλον τρία χρόνια πριν εγκρίθηκαν από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που είχαν προκύψει και πέρασαν βέβαια και από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή ε, αυτή είχε σχέση με τους, ε, ήταν μία από, αυτούς, από αυτές που ασχολούνται με τους ε, χρήστες και εδώ έχουμε μια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία σας δείχνω και η οποία δημοσιεύτηκε ε, μέχρι και ξεκίνησε το 2012, 12 με 14, τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή στο τέλος, στο πέρας της θητείας οι υπηρεσίες αυτές, ε, για να σας το πω πολύ σύντομα, χωρίζονται σε δύο τομείς. Ε, ο πρώτος ε, είναι η πρώην υπηρεσίες επίπτωσης, δηλαδή όλες οι προηγούμενες συζητήσεις, το θέμα της ενασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτά τα προβλήματα και επίσης εδώ δίνει μια αυτόματη έγκριση για τη στήριξη της, ε, ε, των, της, των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής, των πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γίνεται μια διευκρίνηση ε, και μια εξήγηση ε, της συλλογιστικής της Επιτροπής, δηλαδή της συλλογιστικής σύμφωνα με την οποία έγινε ε, ε, έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις. Και γράφονται πολλές σελίδες οι οποίες αποτελούν και ένα είδος οδηγού για τα μέλη όταν χρειάζεται μια αξιολόγηση. Ε, για να ταυτίσουμε τώρα τι επιλογές υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιλέξουμε την, μία, την κάθε επιλογή ξεχωριστά έτσι όπως είναι κατανεμημένες και υπάρχουν και εναλλακτικέ θέσεις για να ε, δοκιμαστεί η ισχύς ή η αδυναμία των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά το επίπεδο των επιπτώσεων και να χαραχτούν ορισμένες γραμμές όπου θα μπορούσαν να ληφθούν και έρευνες σχετικά με αυτές τις δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχικά πριν από δύο χρόνια είχαν ε, υπάρξει όλο και πιο πολλά καινούργια θέματα και όλο και πιο πολύ φόρτος εργασίας με θέματα που προέκυπταν ε, και υπήρχαν ε, συμπληρωματικές πληροφορίες στήριξης, θετική στήριξη και τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής όπου στην έκθεση αυτή είχαμε τα 21 κατατεθειμένες τροπολογίες και όλες αυτές οι αλλαγές είναι γραμμένες, εγγεγραμμένες στην έκθεση πεπραγμένων. Και επίσης για την προστιθέμενη αξία ε, της υπηρεσίας αυτής η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τη Γενική Διεύθυνση να ε, της παράσχει μια στήριξη προστιθέμενης αξίας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ε, έχουμε εδώ αυτήν την εισήγηση με όλες τις καταγραμμένες υπηρεσίες ε, τις, και εδώ έχουμε τις 14 εταιρείες και όλες τις ε, σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 8 έχουμε διεκπαιρεώσει μέχρι στιγμής τέτοιου είδους στηρίξεις προστιθέμενης αξίας και βλέπουμε αν υπάρχει καταρχήν μια νομοθετική πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να παραχθεί αυτή η υπηρεσία και αν μπορεί να γίνει χρήση αυτής της παροχής. Πέρα από αυτό υπάρχει ε, μία έκθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, που αφορά την ανάλυση μίας σειράς δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν έχουν συμπληρωθεί είτε είναι για οικονομικούς είτε για άλλους λόγους, παίρνει διάφορες μορφές και εκεί εγκρίνεται μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ε, η οποία αναλαμβάνεται από τους θεσμούς και έχουμε ε, ένα ε, έχουμε διαφορετική uh, uh, uh, για το κόστος της μη Ευρώπης και νομίζω ότι επίσης μπορούμε να πούμε για μια σειρά θεμάτων ε, οι 25 τομείς πολιτικής όπου παρενέβη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ε, και εξετάζουμε αν εγκρίθηκαν αυτές οι πολιτικές ε, και αν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μιλάμε για ένα τρισεκατομμύριο το χρόνο. Το τρίτο τομέα στον οποίο ε, δρά η γενική μας διεύθυνση είναι οι εργασίες στον τομέα της εφαρμογής και των εργασιών των εμπειρογνωμών ε, σε μια ε, νομοθετική εργασία. Εδώ οι υπηρεσίες έχουν πάρει δύο μορφές εργασίας. Καταρχήν να δώσουν ορισμένες background notes στην Επιτροπή για την εφαρμογή και αυτή η καταγραφή βασίζεται σε ένα μέτρο το οποίο έχει ληφθεί μετά από μία, την έγκριση μιας λευκής βίβλου για ένα πρόγραμμα εργασίας ε, και όπου λέγεται ότι θα, θα καταγράφεται αυτή η σχετική πρωτοβουλία όταν αναλαμβάνεται και παραδείγματος χάρη είχε γίνει αυτό για τους νόμους του copyright το περσινό έτος και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να κατανοήσει ποια ήταν, ε, ποιο ήταν το υπόβαθρο σε ό,τι αφορά όλες τις κρίσεις που υπήρχαν από άλλα θεσμικά όργανα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους θεσμούς. Υπάρχει ανάλυση του Κοινοβουλίου, υπάρχει πληροφόρηση, σχετικές πληροφορίες από όλους τους ετούντες προς το Κοινοβούλιο και τελικά έχουμε... Ε, μια επιτόπια έρευνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλο αυτό το πρόγραμμα κατά την προετοιμασία της Επιτροπής όταν παίρνει στα χέρια της την νομοθετική πρόταση που της έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόλις ξεκινήσαμε αυτή την εργασία... Αυτό το καλοκαίρι και η Επιτροπή είναι ένας από τους πρώτους χρήστες αλλά επίσης όταν λαμβάνεται μια απόφαση αρχής για την εφαρμογή όσον αφορά την οδηγία. Εμεί θα δίναμε παράλληλα τις, τα παράλληλα άλλα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και μια αξιολόγηση εφαρμογής που υπησέρχεται σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς δηλαδή εφαρμόζονται όλα αυτά από νομικής πλευρά σήμερα. Όπως προανέφερα, η Νομική Επιτροπή είναι μείζον πελάτης σε σχέση με αυτά. Μέχρι σήμερα είχαμε αξιολογήσεις ε, τριών ε, τέτοιων υποθέσεων πρόσθετης αξίας ε, και της νομοθετικής διαδικασίας και της, το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Κάναμε δύο εκθέσεις για το κόστος της μη Ευρώπης για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και όσον αφορά το ιδιωτικό δίκτυο και την ελεύθερη κυκλοφορία, όσον αφορά την αποδοχή και διαθεσιμότητα δημοσίων εγγράφων και εργαζόμαστε όσον αφορά την εφαρμογή όσον αφορά την οδηγία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αν επιθυμεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ανασκοπήσει και να δει το τι έγινε στο παρελθόν με πρωτοβουλίες νομοθετικές φυσικά θα μπορούσε αυτό και από πλευρά πλειοψηφία να υποστηριχθεί από την Ολομέλεια. Σε σχέση με θέματα όπου δεν ανταποκρίθηκε η Επιτροπή θετικά μέχρι τώρα και σε σχέση με την έρευνα, για παράδειγμα, και για τις οδικές μεταφορές και τις ε, ε, διαδικασίες. Είναι διάφορα παραδείγματα για τις πρωτοβουλίες που διερευνήθηκαν ε, θέματα κατά το παρελθόν και πρέπει να δούμε ότι υπήρξε καθυστέρηση από πλευρά της Επιτροπής. Όλο το έργο που περιγράφηκε εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και αυτό το ευρύτερο πλαίσιο είναι ο κύκλος πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο να δούμε την πρόταση όταν απορρέει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να δούμε και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Επίσης βλέποντας και και προηγούμενα από πού προέρχεται η πρόταση και ύστερότερα τι γίνεται μετά στην εφαρμογή. Και ουσιαστικά ε, θα ήταν αυτός ο κύκλος που θα πρέπει να ταιριάζει και με τις αξιολογήσεις εξ post για το πώς λειτουργούν τα νομικά αυτά θέματα και ποιες αλλαγές θα επιθυμούσατε να προταθούν για αυτά τα θέματα και ποιες είναι οι μελέτες επιπτώσεων, ποιες επιπτώσεις θα υπήρχαν και ποια θα ήταν τα ωφέλη από πλευρά τέτοιων πρωτοβουλειών. Και υπήρξε μετάθεση προς αυτήν την κατεύθυνση ουσιαστικά κατά τα τελευταία χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και ε, θεσμικά όργανα δραστηριοποιούνται. Εντάσσεται λοιπόν αυτό το έργο σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ σε σχέση με συμπεράσματα υπάρχουν φυσικά σημαντικά θέματα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε αυτές τις εξελίξεις. Στην περίπτωση της ε, εκπροημίου μελέτης επιπτώσεων, εξ άντε, το θέμα που πρέπει να διευθετηθεί δεν μπορεί σε κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή εκπροημίου να αποφασιστεί. Θα μπορούν όμως και θα πρέπει να ενεργοποιούνται περισσότερο οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξετάζοντας τέτοιου είδους θέματα. Κάποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλες δεν είναι τόσο ενθουσιώδεις να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ενδιαφέρον να πει κανείς και να παρατηρήσει ότι όταν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε σχέση με νέο νομοθετικό έργο ή με ένα νέο κύκλο ε, τέτοιων θεμάτων θα μπορούσαν να υπάρξουν νέες ευκαιρίες. Δεύτερον, το θέμα της ε, ε, μελέτης επιπτώσεων και επιτροπολογιών. Και με βάση αυτά, κοινοβουλευτικές επιτροπές προσπαθούν και το θεωρούν κιόλας και επικοδομητικό για τους τριλόγους, τριμερείς διαλόγους όταν οι εισηγητέ και οι σιώδεις εισηγητές ε, εξετάζουν κάποια νομική βάση και γιατί προτείνονται αλλαγές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως θα επιθυμούσαν, θα ήταν ευκταίο να υπήρχαν περισσότερες λεπτομέρειες για ένα τέτοιο νομικό έγγραφο. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όταν είχαμε μια τροπολογία για την ανακύκλωση ε, και σε σχέση με πιο πρόσφατα όσον αφορά τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και γενικότερα επιχειρήσεις όσον αφορά την ε, οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες. Και από πλευρά εισηγητού ε, ενισχύθηκαν κάποιοι τομείς. Στον τομέα της πρόσθετης αξίας, το έργο το οποίο επιτελέσαμε βοηθά να ενισχυθεί το Ευρωκοινοβούλιο έναντι του εκτελεστικού σκέλους, έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με μια ευφιέστερη δραστηριοποίηση για το τι γίνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς δρά. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς, αν δει το πρόγραμμα των 10 σημείων, των κατευθυντήριων γραμμών και προσανατολισμών, υπάρχει υψηλός βαθμός θα έλεγα σύγκλησης σε αυτούς τους τομείς όσον αφορά την ανάλυση, ανάλυση θεμάτων και το έργο που επιτελείται από κοινοβουλευτικές επιτροπές για την πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία. Και τέλος, εξπόστα έργο, δηλαδή αξιολόγηση και επιπτώσεων. Και πάλι εδώ θα θέλαμε να υπήρχε από πλευράς του κενού που παρουσιάζεται σε σχέση με νομικές προτάσεις η κάλυψη των θεμάτων. Υπάρχει μια δυνατότητα, μια πρόπτικη ε, σε σχέση με τις ε, επιλογές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε διευρυμένη υποστήριξη διοικητική για αυτές τις δράσεις ε, με την ανάπτυξη πραγματογνωμοσίας από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης και για την αλλαγή των διαδικαστικών κανόνων και διατάξεων Τώρα, σε σχέση με τις ε, δυνατότητες ε, ε, εφαρμοστικότητας και εφαρμογής μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, αν επιθυμούν, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν με περισσότερη σοβαρότητα τέτοιου είδους θέματα και πρωτοβουλίες. Και προσπαθούμε επίσης να διευρύνουμε, να επεκτείνουμε τις δυνατότητες των υπηρεσιών όσον αφορά για παράδειγμα τη γραμματεία ε, της Επιτροπής ε, ε, εξέταση ρητρών αναθεώρησης σε σχέση με την νομοθεσία για τα όσα εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με την επισκόπηση, η αναθεώρηση, η αξιολόγηση εδώ διοργανώ, διοργανώνεται από την, ε, από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή μια τέτοια δυνατότητα για την ex post ανάλυση. Επαρκούμε σε αυτές τις παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πολύ σαφές, ε, σαφής η ανακοίνωσή σας, πολύ συγκεκριμένη, σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να λάβει το λόγο, να ζητήσει κάποια εξήγηση, παρακαλώ κύριε Λιμπέα. και μετά ναι. Η κυρία Νίμπλερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον κύριο Τίσντελ και τους συναδέλφους και συναδέλφους γυναίκες και άνδρες. Νομίζω ότι οι δομές που δημιουργήθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε το πολιτικό μας έργο ουσιοδός να μπορέσει να υποστηριχθεί είναι μοναδικό αυτό το έργο και θέλω και πάλι να ευχαριστήσω Μία έκθεση κοινοβουλευτική που από πλευράς της ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε δεν το είχαμε ξαναζήσει μέσα σε ένα χρόνο να εφαρμόζεται τόσο, με τόσο ουσιώδη τρόπο και τόσο αποτελεσματικά όπως από τη δική σας μονάδα. Και τώρα με την μετεξέλιξη της, του έργου σας για το κόστος της μη υλοποίησης της Ευρώπης, το κόστος της απουσίας της Ευρώπης και όλων των λοιπόν θεμάτων βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά αυτά τα θέματα που αναλύσατε και είναι πολύ επιτυχές το έργο σας και θέλω να το εκφράσω αυτό και θα χαιρόμουν αν θα, μπορούσαμε να συνεχισ... αν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η πορεία όπως την ακολουθήσατε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αναφέρεται συγκεκριμένα στο ότι έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο τώρα πλέον και πολλοί συνάδελφοι για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιούνται ως ευρωβουλευτές. Εσείς τι κάνετε, πάτε και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και μεριμνάτε ώστε αυτά τα μέσα τα οποία θα μπορούν να διατεθούν στους ευρωβουλευτές και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές να διατίθενται σε αυτούς. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, τέτοια ζήτηση και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό το έργο το δικό σας ώστε από κοινού αυτή η πραγματογνωμοσύνη και η τεχνογνωσία να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πλευράς μας. Και η δεύτερη ερώτηση είναι περισσότερο πολιτική. Είχαμε τις ακροάσεις των επιτρόπων, γυναικών και ανδρών, για την Επιτροπή τον, τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουμε και έναν αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμαν, που είναι και αρμόδιος για τα θέματα απελευθέρωσης αγορών, αντιμετώπιση του γραφειοκρατικού βάρους και θα είναι της γραφειοκρατίας και θα είναι και αρμόδιος για θέματα επικουρικότητας και θα ήθελα να ζητήσω από αυτή την ε, ισόρροπη δράση πώς ε, θα μπορέσουν να αξιολογηθούν αυτά από την Επιτροπή. Είχαμε ζητήσει να υπάρξει μια ανεξάρτητη υπηρεσία, ένας ανεξάρτητος φορέας που θα μπορεί να, επικουρεί, να ε, συνδράμει τα θεσμικά όργανα και που ίσως και από τον αντιπρόεδρο αυτό θα μπορούσε μια τέτοια ανεξάρτητη μονάδα να δράσει και να βοηθήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ήθελα να πω να ξέρουμε ότι όλα τα κοινοβούλια του κόσμου έχουν τέτοιες υπηρεσίες επαλήθευσης, ελέγχου, επιθεώρησης, στήριξης πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι πολυτέλεια, πρόκειται για μία πρόληψη προβλημάτων. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός και να γίνεται τακτικά μία, ένας έλεγχος ποιότητας. Παρακαλώ κυρία μου, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω πόσο εκτιμώ αυτού του τύπου την υπηρεσία που έχουμε στη διάθεσή μας που καταρτίστηκε πρόσφατα και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτή την επιθεώρηση η οποία γίνεται. Υπάρχουν ορισμένες, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, οι προϋποθέσεις οι οποίες δεν πληρούνται και ότι χρησιμοποιείται η υπηρεσία σας όταν ε, καλείτε να καλύψει ορισμένους τομείς όπου υπάρχουν κενά ε, στον τομέα της παροχής αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλώ. Κύριε Τισδέλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για να απαντήσω τώρα με τη σειρά της ερωτήσεις, καταρχήν βεβαίως κάθε επιτροπή θα μπορούσε, να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, κάθε, κάθε επιτροπή θα μπορούσε να έχει το δικαίωμα σε μια τέτοιου είδους παρουσίαση, θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό και, το, και έλεγξα τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει παρουσιάσεις σε εννιά κοινοβουλευτικές επιτροπές και έχουμε ε, συντονισμό ε, εισηγητών και σκιωδών εισηγητών σε οχτώ επιτροπές. Βεβαίως κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου παρουσιάστηκαν και άλλες πολλές έρευνες και ε, νομίζω ότι μπορούμε ε, να χρησιμοποιηθούμε σωστά για να καλύψουμε ένα ολόκληρο φάσμα και θα χαιρετίζαμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και θα παρουσιάσαμε το έργο μας όσο πιο πλατιά γίνεται. Τώρα υπάρχει ένα πιο πολιτικό ερώτημα το οποίο αφορά τον νέο αντιπρόεδρο ε, που, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι δική μου υπόθεση βεβαίως ούτε της δικής μου εμβέλειας να εκφέρω κάποια κρίση να κάνω κάποια αξιολόγηση για αυτό το θέμα ξέρουμε όμως ότι υπάρχει μια αλλαγή στο επίπεδο της πολιτικής χρειάζεται μια εμπειρογνωμοσύνη και μια στήριξη σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης ε, και γι' αυτό λέγεται περισσότερη ρύθμιση ε, με έναν πιο κομψό τρόπο τρόπο αυτού του είδους ο περιορισμός και αυτού του είδους η στήριξη μέσα από περισσότερες εμπειρογνωμοσύνες και υπάρχει μεγάλη προτεραιότητα για την ώρα που δίδεται σε αυτή την ανάγκη. Ε, οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ καλές στην αρχή ήπιες όταν ε, ασχοληθήκαμε με διάφορα πεδία εργασία υπήρχε στην αρχή ο φόβο και η ανησυχία να υπάρξει, να μήπω υπάρξει κάποια αντιπαράθεση, κάποια προστριβή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τελικά είδαμε τους, ότι οι γραμματεί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανακάλυψαν ότι ε, είχαμε αυτήν την υπηρεσία, προσπαθήσαμε να του βοηθήσουμε και του δείξαμε ότι υπάρχουν διάφορε ε, κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορούσαμε να δράσουμε. Ένα από τα προβλήματα αυτής της στήριξης ιστορικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι εκεί υπάρχουν διάφορες γενικές διευθύνσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και η Γενική Γραμματεία προσπάθησε για πάρα πολλά χρόνια με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία μέσα στα χρόνια να τα εναρμονίσει όλα αυτά και ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρθηκε έντονα για αυτό το θέμα και ζήτησε μια στήριξη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο για την άποψή μας ήταν πάρα πολύ θετικό. Και επίσης υπάρχει το ερώτημα του αν ε, αυτή η στήριξη ε, της, ε, των επιπτώσεων είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με το έργο του, με το, με το τι ζητάει το Κοινοβούλιο στήριξη ε, και τελικά όταν ξεκινήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίσταζε πάρα πολύ για όλες αυτές τις διαδικασίες ε, και δεν έδειξε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. δεν είχε ενδιαφέρον. Στην αρχή ε, ήταν έτσι τα πράγματα. Στη συνέχεια και πριν από το τελικό κείμενο υπήρχε μια, υπήρξε μια ιστορικού χαρακτήρα εισήγηση η οποία εξηγούσε τα πράγματα και η οποία επαναδιατύπωσε αν θέλετε όλα τα θέματα των μελετών επιπτώσεων και των αξιατικών αξιολογήσεων και τελικά το Κοινοβούλιο ε, χρησιμοποίησε αυτές τις ε, μελέτες επιπτώσεων στην Επιτροπή δεν δόθηκαν, δεν παρασχέθηκαν σχετικές άδειες ε, παραδείγματος χάρη για ότι μπορεί να μην ε, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια μελέτη επιπτώσεων. Είναι μια εργασία που την είχαμε ε, ε, παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο και υπήρξε και ένα σχετικό ψήφισμα από ό,τι θυμάμαι. Βεβαίως αν δεν έχουμε λάβει κάποια στιγμή εντελώς διαφορετικές εντολές θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως δουλεύαμε και βασιζόμενοι στις αναλύσεις μας τελικά υπάρχει μια προοπτική διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Η κυρία ε, Τόπιν με ρώτησε για την ενημέρωση όλων αυτών των κειμένων και των εισηγήσεων. Κάθε πέντε χρόνια έχει αποφασιστεί να γίνεται μια τέτοια ενημέρωση, 2014 με πίσω 2009 και δίδονται βεβαίως πολλές πληροφορίες σε αυτά τα έγγραφα. Ε, όχι όμως ικανές, θα, θα χρειαζόταν κάτι περισσότερο και υπάρχουν ορισμένες προτάσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί κάποιες ανακρίβειες. Πρέπει όμως η σχετική υπηρεσία να είναι σε θέση όπως και είναι να εξετάζει αναδρομικά όλα αυτά τα θέματα και να βλέπει τι είδους απαντήσεις δόθηκαν σε ορισμένους τομείς ε, όπου έχει γίνει σχετική, έχει συνταχθεί η σχετική νομοθεσία, η σχετική νομοθετική πρόταση και ε, μέσα στην Ευρώπη είναι κάτι αυτό το οποίο συμβαίνει συχνά και χρειάζεται τέτοιου είδου στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τίσδελ θέλει κανείς κάποια άλλη πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω εάν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όταν είναι οι εισηγητές, οι σκιώδεις εισηγητές μπορούν να προσφύγουν σε εσά όταν έχουν, θέλουν στοιχεία έρευνας και στήριξη. Έχω μια... Ε, απάντηση γι' αυτό, αλλά υπάρχει η γενική εργασία καταρχήν πρέπει να πω ε, που και η εργασία που γίνεται για λογαριασμό ατομικών μελών ε, που είναι μια συγκεκριμένη υπηρεσία ε, η οποία αφιερώνεται σε αυτά τα θέματα. Όταν γίνεται λοιπόν μια αξιολόγηση, μια μελέτη επιπτώσεων, πάντα η είναι δυνατόν να γίνει και να υπάρξει μια ενημέρωση και ένα μέλος της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει μια ενημέρωση της μελέτης επιπτώσεων Βεβαίως δεν θα, δεν θα ήμασταν στη διάθεση ενός μόνο κράτους μέλους, αλλά όλες οι δημοσιεύσεις μας και όλες οι μελέτες μας είναι πάρα έχουν μεγάλο εύρος και καλύπτουν ε, πάρα πολλά θέματα πάνω στα οποία εργάζονται οι επιτροπές και η δική σας επιτροπή συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ και το νομικό σύμβουλο και την ομάδα του που μας εξήγησαν τη λειτουργία τους. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω να εκτιμάτε όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή σας ως πληροφόρηση και ως αξιολόγηση των εργασιών. Θα περάσουμε τώρα. Θα περάσουμε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης. Παρουσίαση της έκθεσης του κυρίου Φως αλλά αντικαθίσταται από έναν άλλο συνάδελφο, ο κύριος Φως. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ψηφίσουμε για το θέμα της νομικής βάσης σύντομα. Και αυτό επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη σύμβαση για το εμπόριο της ε, άγριας ε, χλωρίδας και πανίδας προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών ζητήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, να ασχοληθεί η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο και να γνωμοδοτήσει σε σχέση με τα στοιχεία της πρότασης. Υπάρχουν τρία στοιχεία σε σχέση με την νομική βάση. Το άρθρο της Συνθήκης 192 νομική βάση για το περιβάλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά έχουμε και το 207 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον έχουμε και το άρθρο 218 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις διαδικασίες και διεργασίες και όσον αφορά την νομική βάση για την σύναψη διεθνών συμφωνιών ε, ε, για τα θέματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Ευρωκοινοβούλιο και σε σχέση με το 207 για το αίτημα συνένεσης από πλευράς του ε, Συμβουλίου προς το Κοινοβούλιο στην πρώτη σύμβαση που πρέπει να ζητείτε η προστασία, να διασφαλίζεται η προστασία αυτή με καλύτερες εμπορικές συμφωνίες η ένταξη σε αυτή τη ε, σύμβαση, σε αυτή τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εντάσσεται σε αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές και να καλύπτονται όλες όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται διαδικαστικά και σε σχέση με διεθνείς συμφωνίες για την προστασία αυτών των ε, ειδών, καθώς επίσης ε, και οι πτυχές εμπορίου. Αυτή είναι η πρόταση η οποία υποβάλλεται από τον άξερφος εισηγητή και μου ζήτησε να σας διαβιβάσω αυτά τα στοιχεία πληροφοριακά προς εμάς και επίσης προστίθεται ότι σε σχέση με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τη γνωμοδότηση αυτή η άποψη ευθυγραμμίζεται πολύ με τα στοιχεία τα οποία σας έδωσα και σας ευχαριστώ. Σα euh, Σας ευχαριστώ. Αναπληρώσατε επάξια τον συνάδελφο Φως. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρατήρηση πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Δεν νομίζω. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν της εκθέσεως Φως. Ποιοι είναι υπέρ. Κρατήστε ψηλά τα χέρια σας παρακαλώ γιατί πρέπει να καταμετρηθούν. είναι κατά. Αποχές. Καμία αποχή. 15 υπέρ, 6 κατά. Έχει εξασφαλιστεί και η απαρτία. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι το 8. Θα πρέπει εδώ ε, για την έκθεση Σβόμποτα, για την επιλογή δικαστικής αρχής, η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 20 Οκτωβρίου 12η μεσημβρινή. Μιλάμε για την έκθεση Σβόμποντα. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 8, ειδικό πρωτόκολλο για, για την κινούμενο σιδηροδρομικό εξοπλισμό. Το λόγο έχει η κυρία Χάουταλα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό είναι κληρονομιά από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το Κοινοβούλιο τώρα ζητείται να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του στη διαδικασία του Συμβουλίου για το πρωτόκολλο κινητού σιωδρομικού υλικού. Είναι το λεγόμενο Rail Protocol, εν δεν είναι περίπλοκο το θέμα αυτό, δεν παρουσιάζει προβλήματα, αλλά παρατηρώ εδώ ότι έχει υπάρξει μια κάποια καθυστέρηση από τότε που το Συμβούλιο υπέγραψε αυτό το Διεθνές Πρωτόκολλο από τις 10 Δεκεμβρίου του 2009. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να δημοσιεύσει το Συμβούλιο την πρότασή του. Ίσως κάποιοι εμπλεκόμενοι, κάποια εμπλεκόμενε κάποιες ε, εμπλεκόμενες πλευρές λοιπόν ε, προκάλεσαν αυτή την καθυστέρηση. Συνδέεται με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Στόχος είναι να γίνουν οι επενδύσεις στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους περισσότερο ελκυστικοί, ελκυστικές οι επενδύσεις. Στόχος του πρωτοκόλλου είναι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης κινητών εξοπλισμών στον τομέα του σιδηροδρόμου υψηλής ποιότητας. Είναι κάτι το οποίο θα έχει σαν στόχο επίσης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα. Η πρόταση του Συμβουλίου παρατηρεί ότι κάποια άρθρα του πρωτοκόλλου συνδέονται με θέματα επιλεκτικών ε, προτιμήσεων σε τομείς όμως όπου έχει ήδη πάρει αποφάσεις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι γύρω από το θέμα αυτό. Απλά θα πρέπει να δώσουμε μια σύμφωνη γνώμη στην απόφαση του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κέστερ. Ως κοιόδη εισηγητής για τους Σοσιαλδημοκράτες μπορώ να πω ότι συμφωνούμε με αυτά τα οποία πρότεινε η κυρία Χαούταλα. Είναι σκόπιμο αυτό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πιστωτών και μπορεί να συνεισφέρει να προαχθούν οι επενδύσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τους σιδηροδρόμους και η πτυχή της αηφορίας ε, ενισχύεται και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι το σκόπιμο και κάτι το οποίο έχει νόημα και θα το υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Κυρία Χάουταλα, μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις προθεσμίες για την κατάθεση των τροπολογιών. Δεν γνωρίζω τις προθεσμίες, λέει η κυρία Χάτουλα, ίσως η γραμματεία. Και η γραμματεία δεν έχει γνώση αυτών των προθεσμίων των χρονικών. Θα σας ενημερώσουμε γραπτά για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάουταλα, η πρόταση από την Γραμματεία είναι 24 Οκτωβρίου. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 24η. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Ε, περνάμε στο επόμενο θέμα. Η κυρία Λεγκρίπη είναι η συγγήτρια, δεν υπαρχει καποιο προβλημα εδω περναμε στο φτάσει ακόμα. Ίσως θα περάσουμε στο μεθεπόμενο θέμα. Επικουρικότητα λοιπόν. Το λόγο έχει η κυρία Ντελβοστέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια οδηγία η οποία τροπολογεί έξι διαφορετικές οδηγίες παλαιότερες για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις χωματερές, την ανακύκλωση συσσωρευτών, μπαταριών κτλ. Η επί της ουσίας αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος βέβαια. Έχουμε ήδη λάβει δηλαδή, μια αιτιολογημένη γνώμη από την Αυστρία που λέγει ότι το θέμα αυτό είναι περιφερειακό θέμα ε, και εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε να δούμε αν υπάρχει επί τη βάση της αρχής της επικορικότητας ε, ε, δυνατότητα παρέμβασης σε επίπεδο κοινοτικό. Απαντώντας στην Αυστρία μπορούμε να πούμε ότι η οδηγία αυτή τροπολογεί τις ισχύουσες οδηγίες. Δεν ορίζει νέους κανόνες, Θέτει όμως ορισμένους στόχους οι οποίοι είναι κοινοί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σύμφωνα με τις οποίες κάθε χώρα και κάθε περιφέρεια διαχειρίζεται τα απόβλητα αλλά με κοινού στόχους. Δεν υπάρχει λόγος παρέμβασης λοιπόν εδώ και δεν υπάρχει λόγος να επιστήσουμε την κίτρινη κάρτα Ας αφήσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος να εργαστεί κανονικά σε σχέση με τη συγκεκριμένη οδηγία. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρέμβαση. Όχι. Καλώς. Προχωράμε αρκετά γρήγορα και θα εξαντλήσουμε την ημερήσια διάταξη πριν μας εξαντλήσει αυτή. Περνάμε λοιπόν στο 11. Φτάσαμε στο σημείο 11 Ίσως να χρειαστεί να διακόψουμε για λίγα λεπτά μάλλον λέει ο πρόεδρος ώσπου να φτάσει η κυρία Λεγκρίπ. Είναι 4 και 20, σας προτείνω παρακαλώ να βρεθούμε στα 10 λεπτά. Ίσως, συγγνώμη, ίσως να ακούσουμε την παρουσίαση ε, της νομικής υπηρεσίας όσο παραμένουμε στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα αποφασίσω για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 14ης Ιουνίου για την υπόθεση Αταλάντα Μαωρίσιους. Θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί αυτή είναι η διαδικαστική γλώσσα η οποία επελέγει από το Κοινοβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η περίπτωση Αταλάντα Μωρίσιος είναι ένα σημαντικό βήμα για την δημοκρατική εξέταση της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η περίπτωση αφορά την ρήτρα που αποκοινούμε τα δικαιώματα του Ευρωκοινοβουλίου για να εγκρίνει ή απορρίπτει διεθνείς συμφωνίες υπό το αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και το δικαίωμα του Ευρωκοινοβουλίου άμεσα να πληροφορείται άμεσα σε όλες τις φάσεις για τις διαδικασίες υπό το άρθρο 218 παράγραφο 6 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε πέντε κράτη-μέλη υπέρ του Συμβουλίου ζητήθηκε σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή. Μια στιγμή αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Ευχαριστώ λοιπόν γιατί θα είναι πιο χρήσιμο τώρα αν μπορείτε ναι, για να μην υπάρχει λοιπόν σύγχυση, ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου σε σχέση με τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για την μεταφορά όσον αφορά πειρατών και περιουσιακών στοιχείων που είχαν κατασχεθεί σε σχέση και με τις ε, δράσεις ε, ύποπτες για πειρατεία. Το Κοινοβούλιο βασίστηκε σε δύο ε, περιπτώσεις την παραβίαση της αρχής της αμοιβαιότητας και έλλειψη ή ελλειπή πληροφόρηση από το Συμβούλιο ουσιαστικά το, το Κοινοβούλιο είδε να, ότι παραβιάζεται η συνθήκη κατάφορα. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι έγινε αυτή η συμφωνία από το Συμβούλιο με βάση το αποκλειστικά το άρθρο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άρθρο το οποίο αφορά την εξωτερική πολιτική, χωρίς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή χωρίς να ζητηθεί και η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θεώρησε ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά επίσης αφορούσε τον κοινό χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ε, δημοκρατίας. Και έτσι λοιπόν θεώρησε ότι θα έπρεπε να εφαρμόζονται αυτές οι διαδικασίες αναλύοντας ε, τα όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο, θεώρησε ότι αυτή η δυνατότητα δεν προβλέπει μόνο μία αποκλειστική ερμηνεία αυτή η περίπτωση και θεωρήθηκε ότι ο όρος αποκλειστικός στην ε, ε, διατύπωση αυτή δεν μπορεί μονομερός να ερμηνεύεται αλλά είναι αναγκαίο να εξεταστεί σύμφωνα με, τις, με τους στόχους και τις περιπτώσεις μέσα στις οποίες και στους οποίους ε, αναπτύσσεται αυτή η δράση. Και γι' αυτό <clears throat> σε σχέση με την ανάλυση και ε, των στοιχείων αυτής της συμφωνίας το δικαστήριο φαίνεται ότι ε, θεωρεί ότι υπήρξε μόνο μία αποκλειστική ερμηνεία. Γι' αυτό τον λόγο απορρίφθηκε λοιπόν η πρώτη προσφυγή. Στην δεύτερη προσφυγή ε, ισχυρίστηκε το Κοινοβούλιο ότι είχε παραβιαστεί το άρθρο 218 της, ε, συμφων... συνθήκης γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση σε σχέση με αυτή τη συμφωνία και την ανάπτυξή της ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά μόνο τρεις μήνες μετά την και δημοσίευση αυτής της συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αντίθετα σε σχέση με τα επιχειρήματα που παρουσιάζει το Συμβούλιο και τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 218 αφοράται εδώ. Και θεώρησε το ε, Συμβούλιο ότι το άρθρο 210 μπορεί να εφαρμόζεται, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις ε, που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική. Έτσι λοιπόν αυτή η διάταξη για την ε, συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης πρέπει να εφαρμόζεται για την κοινή εξωτερική πολιτική. Ωστόσο όμως σε σχέση με την ε, ε, συμφωνία αυτή παρόλες τις ε, σαφείς διατυπώσεις το Συμβούλιο δεν θεώρησε ότι υποχρεούτο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και σε σχέση με την φάση σύναψης, ε, ολοκλήρωσης της συμφωνίας ε, δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο και έτσι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και ούτε ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου, η συνένεσή του. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με το άρθρο 218 218-10 δεν υλοποιήθηκαν τα όσα προβλεπόνσαν Ωστόσο όμως ε, το δικαστήριο δεν ακολούθησε την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα ενώ γενικά ακολουθεί τις συστάσεις του. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με τις ε, ενστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρήθηκαν ότι ευσταθούσαν και γι' αυτό σε σχέση με τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ Μαυρικίου ακυρώθηκε. Και πρώτα απ' όλα σε σχέση με το αποδεκτό αυτή της διαδικασίας θεώρησε το ε, δικαστήριο ότι σε σχέση με το άρθρο 218 πρέπει να εφαρμόζεται αυτό γενικά και γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες ε, που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς ε, δραστηριοτήτων της καθώς επίσης και στην κοινή εξωτερική πολιτική και το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει σε σχέση με τη δεύτερη προσφυγή, το δικαστήριο σε σχέση με τη δεύτερη προσφυγή με σαφήνεια δηλώνει ότι καθώς το Συμβούλιο δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο όπως θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφο 10 υπήρξε παραβίαση των προβλέψεων της συνθήκης. Το δικαστήριο τόνισε ότι οι διατάξεις που προβλέπονται αποτελούν ισχυρές και ε, αναγκαίες συνθήκες και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με το άρθρο 263 της συνθήκης. Και αυτή η παραβίαση οδηγεί στο να μην μπορεί να ισχύει μια τέτοια συμφωνία. Σύμφωνα με το δικαστήριο η παραβίαση του δικαιώματος ενημέρωσης και πληροφόρησης του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με σημαντικά θέματα αυτής της συμφωνίας, αυτής της συνθήκης παραβιάζει τα δικαιώματα του ε, Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και γι' αυτό είναι παραβίαση μιας σημαντικής προϋπόθεσης. Και έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει άμεσα να ενημερώνεται, πλήρως να ενημερώνεται για, την φάση και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και σε σχέση με τις ε, διατάξεις ε, ε, διαπραγμάτευσης και μάλιστα υπό την προοπτική συμφωνίας, σύναψης μιας συμφωνίας καθώς επίσης και για όλες τις ε, προτάσεις ε, που θα πρέπει να οδηγούν στο να ακυρώνονται τέτοιου είδους ε, συμφωνίες. Αυτό ισχύει σε όλες, για όλες τις συμφωνίες και για την είπα το εκπρόσωπο και το Συμβούλιο επειδή είναι μια πολύ σημαντική ε, αναγκαία συνθήκη για τέτοιου είδους συμφωνίες. Αν δεν γίνονται σεβαστές αυτές οι διατάξεις τότε είναι άκυρες οι πράξεις ε, του Συμβουλίου και γι' αυτό θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο συμφωνίας του 2010 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου ιδιαίτερα όσον αφορά την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τακτά διαστήματα να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λαμβάνεται υπόψη πάντα το δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Επίσης η ύπατος εκπρόσωπος, η ύπατη εκπρόσωπος έκανε μια ε, τοποθέτηση σε σχέση με τα, τις διατάξεις αυτές για ένα πλαίσιο συμφωνίας ε, και τα θέματα τα οποία θα εντάσσονται σε τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες. Εν τέλει, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο hm, το 2014 τον Μάρτιο ολοκλήρωσαν μια διοργανική συμφωνία σε σχέση με την ε, ε, ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με απόρριτα ή ε, διαβαθμισμένα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το Συμβούλιο σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σε σχέση με την συμφωνία αυτή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τανζανία για τους όρους μεταφοράς υπόπτων πειραντίας σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο στις 28 Μαΐου 2014 είχε υποβληθεί. Φυσικά αναμένουμε την ε, γραπτή διαδικασία και σε αυτή την περίπτωση έχουμε πάλι δύο πρόσφυγες. Το ένα είναι το δικαίωμα άμεσα να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, το Κοινοβούλιο για τέτοιου είδους θέματα και το άλλο αφορά το δικαίωμα της ε, ε, εφαρμογής της ορθής νομικής βάσης. Αυτά εν συντομία. Είμαστε στη διάθεσή σας αν υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια ή απορίες. Και φυσικά θα μπορούσα να προσπαθήσω να απαντήσω σε οτιδήποτε προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλετε μήπως να παρέμβετε. Φαίνεται ότι οι εξηγήσει ήταν τόσο σαφείς που δεν υπάρχουν ερωτήσει, Η κυρία Χάουταλα, η οποία προσέχει τα πάντα σε κάθε περίπτωση. Λυπάμαι ε, που σήμερα μιλάω τόσο, παίρνω τόσο συχνά το λόγο. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξήγηση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τις νομικές υπηρεσίες το εξής. Ε, υπάρχουν νομικές υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν, για τις οποίες προκύπτουν κάποιες, κάποια συμπεράσματα τα οποία συνάγει η νομική υπηρεσία με την, ε, σχετικά με την ε, θέση του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να είναι πλήρως πληροφορημένο για όλα τα διοικητικά και πολιτικά θέματα των εθνικών διοικήσεων και ότι έχει αυτό το δικαίωμα. Τώρα το ερώτημα το δεύτερο είναι το πλαίσιο, η συμφωνία πλαίσιο του 2010 πρέπει να επανεξεταστεί, πρέπει να ε, εξεταστεί η διοργανική συμφωνία του 2014 που αναφέρατε σε σχέση με αυτή την απόφαση. Παρακαλώ. Ε, ε ευχαριστώ. Για το δεύτερο ερώτημα θα έλεγα ότι εξετάζει, ε, είναι μια πολιτική επιλογή και από αυτό εξαρτάται. Για το πρώτο βεβαίως θα πω ναι ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η διοργανική συμφωνία με το Συμβούλιο γιατί υπό το φως αυτής της απόφασης φαίνεται αν πρέπει να γίνει κάτι σε σχέση με όλες τις συμφωνίες που έχουν συναυθεί σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, κοινή ε, στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής. Για το τρίτο ερώτημα σχετικά με αυτό θα ήθελα να πω ότι όπως υπογράμμισα μέχρι στιγμής το Συμβούλιο δεν έχει κάνει κανένα βήμα σε σχέση με την εφαρμογή της, ε, των αποφάσεων του, της απόφασης αυτής του δικαστηρίου. Οπότε περιμένουμε. Περιμένουμε μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου, τόσο ώστε να κάνουμε το απαραίτητο βήμα προς μια απόφαση, διότι πριν από την απόφαση που εγκρίνει το Συμβούλιο για την σύναψη αυτής της συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας του Μαυρικίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή είναι άκυρη. Έχει κηρυχθεί από το δικαστήριο ως άκυρη και οπότε αυτό ε, είχε, είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί από όλα τα αφορόμενα μέρη και η πρόταση αυτή ε, ακολουθεί ε, την θέση όλων των αφορομένων μερών. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό την παρούσα στιγμή να υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία του Συμβουλίου τους ώστε να αντικατασταθεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου με μια άλλη και να είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις για την σύναψη της ενδεχόμενης μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας με άλλα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Πήρατε ό,τι πληροφορία θέλατε κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ λοιπόν. Τελειώσαμε νομίζω μετά από αυτά και πριν εξαντληθούμε πλήρως θα επανέλθουμε στα προηγούμενα. Ε, στο σημείο 9 της ε, ημερήσιας διάταξης ε, οπότε ήρθε η κυρία από την άλλη επιτροπή που, όπου ήταν προηγουμένω, Θέλατε κάτι να πείτε παρακαλώ μου κάνετε ένα σινιάλο ή ένα σινιάλο σε κάποιον συνάδελφο. Α έρθουμε στο σημείο 9 λοιπόν της ημερήσιας διάταξης που αφορά την προστασία των εμπορικών γνώσεων, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών υποθέσεων όπως την ονομάζουμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή βιομηχανία ε, των άλλων υπήρων και των άλλων ε, ε, οντοτήτων. Παρακαλώ. Συνεχίζουμε τη διαδικασία μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από όλα τα μέλη της Νομικής Επιτροπής για την καθυστέρηση με την οποία ήρθα εδώ. Πραγματικά είχα, έχουμε καμιά φορά προγράμματα που επικαλύπτονται και γι' αυτό. Ε, πριν από λίγο άκουσα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσίασε το θέμα το σχετικό με την οδηγία που μας απασχολεί σήμερα και θα ήθελα πριν από όλα να αντιδράσω σε αυτήν την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ε, διαδικασία παρακολούθησης του κειμένου. Σήμερα ξεκινάμε στη, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τις εργασίες και τη συζήτησή μας πάνω σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι νομοθετικά σημαντικό. Ε, προηγουμένως είπε η Επιτροπή ότι κάπως είχαμε θίξει αρχικά το θέμα ε, εξαπλώνων ήχων, όμως τώρα ένα από τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που δεν είναι πια εδώ, ε, η κυρία Μαριά Τικαλό, η οποία ήταν τότε η συγγήτρια, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια σειρά από άξονες, υποθέσεις ε, και πραγματικά θέλω να τις αποτείνω έναν φιλικό χαιρετισμό με αυτή την ευκαιρία. Έχουμε λοιπόν αυτό το κείμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις οικονομικές ε, επιδόσεις και είναι σημαντικό ότι φαίνεται μέσα σε αυτό το κείμενο μια πραγματική ανάγκη επαλήθευσης. Υπάρχει η πραγματική αυτή ανάγκη ε, ε, για να μπορέσει να εξεταστεί κάτι το οποίο το ακούμε στις προεκλογικές εκσταθίες πάρα πολύ συχνά ε, ακούμε τους ε, συμπολίτες μας να κατηγορούν την αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρώπη γενικότερα ότι νομοθετεί υπερβολικά, ότι νομοθετεί σε τομείς που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας. Εν πάση περιπτώσει εδώ διαπιστώνουμε ότι η προστασία της τεχνογνωσίας, των διαφόρων τεχνογνωσιών είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν πολλοί εταίροι που εκδηλώνουν την πραγματική ανάγκη κοινή νομοθεσίας και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, έχουμε πληροφορίες τις οποίες εισάγουμε ε, οι μεν και οι δε σε αυτήν την κοινή υπόθεση ώστε να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας, στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αφήσει ημιτελή αυτή τη διαδικασία που αφορά την ανανέωση της Ευρώπης μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και ε, η υπόθεση αυτή έτσι όπως έχει καθοριστεί είναι, αποτελεί μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ε, μυστικά εμπιστευτικές υποθέσεις εμπορικές τις οποίες, οι οποίες τους δίνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εμπορικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Αυτή η τεχνογνωσία η μυστική είναι ένα είδος κεφαλαίου ε, διανοητικού που, που είναι άειλο πάρα πολύ συχνά και το οποίο προσελκύει ε, τους αντιπάλους και πρέπει να προστατευτεί. Είναι πολύ βασικό να δώσουμε εγγύηση ε, νομική έναντι όλων των προσπαθειών ε, που γίνονται παράνομα από, ε, για την απόκτηση αυτής της τεχνογνωσίας την παράνομη ε, και βεβαίως πρέπει να περιοριστούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσουμε αυτές τις προσβάσεις και να τιμωρήσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή την παράνομη επέμβαση. Χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των τεχνογνωσιών, των εμπιστευτικών ε, υποθέσεων. Αυτό έχει δύο επιπτώσεις, διπλές μάλλον, ε, για την καινοτομία. Καταρχήν δεν υπάρχει σε ορισμένα κράτη-μέλη εγγύηση, προστασία του μυστικού, ε, του εμπιστευτικού χαρακτήρα. Υπάρχει για τους επιχειρηματίες μια νομική κάλυψη και μια ασφάλεια η οποία χρειάζεται να αυξηθεί σε σχέση με όλες τις νομοθεσίες οι οποίες δεν είναι καθόλου ευθυγραμμισμένες μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην εσωτερική αγορά λοιπόν αυτό είναι ένας περιορισμός για τις συνεργασίες και ειδικά για τις διαμεθοριακές συνεργασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εδώ και μερικούς μήνες προσπάθησε κατά κάποιον τρόπο να προσεγγίσει αυτές τις ε, νομοθεσίες και δίνει ένα είδος εργαλείο, μια σειρά από εργαλεία σημαντικά για να υπάρξει μια ασφάλεια νομική. Και εδώ έχετε τα σχέδια των κειμένων που αποτελούν μια πλατφόρμα εργασιακή, μια βάση ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την κοινή μας εργασία, για την εκπόνησή της. Είναι μια βάση πολύ ενδιαφέρουσα, επαναλαμβάνω, και πρέπει να την αναγνωρίσουμε ως τέτοια και την αναγνωρίζει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη της Γενικής Διεύθυνσης των Επιτροπών Μπαρνιέ και το γραφείο του που μας έχει δώσει αυτές τις, ε, αυτά τα κείμενα, αυτές τις εισηγήσεις τεράστιας ποιότητας. Αυτό το κείμενο λοιπόν το οποίο ε, προσπαθούμε να ε, τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε έχει επίπτωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας που είναι και ο κύριος ιστός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ε, και πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληροφορίες, τεχνογνωσίες που είναι βασικές για την επιβίωσή τους την ίδια, επιβίωση της κάθε επιχείρησης, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, η προστασία των γνώσεων, των μυστικών για να υπάρχει αποδοτικότητα και ε, ανταγωνιστικότητα για τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στις επιχειρήσεις αυτές. Μπορούμε να διαπιστώσουμε σε ό,τι αφορά την ε, διαπίστωση του know-how των ε, τεχνογνωσιών ότι χρειάζεται, υπάρχει αυτή η πιστοποίηση που είναι μια επιπρόσθετη σιγουριά και ασφάλεια το να υπάρχει λοιπόν ένα μυστικό, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας μιας πληροφορίας και να προστατεύεται είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ξεκινάει κανείς διαδικασίες χρονοβόρες και πολύ ε, ακριβές. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ευρωπαϊκό ε, ε, πτυχίο ευρεσιτεχνία, πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας που μπορεί να δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια η διαδικασία είναι μακρότατη, χρονοβόρα, ε, δεν θα περατωθεί αύριο, αλλά πάρα πολλοί εταίροι ε, δείχνουν ενδιαφέρον και στο επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στις μεγαλύτερε επιχειρήσει, ε, δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον για αυτό το πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας για, για πολύ λεπτές υποθέσεις το σχέδιο οδηγίας αυτό διασταυρώνει διάφορες ε, προβληματικές πολύ ευαίσθητες όπως είπα και που αγγίζουν θεμελιακά διακυβεύματα ε, για το θέμα της ε, χρησιμοποίησης της σωστής της, της πληροφόρησης και το θέμα του ποιος κυριαρχεί την πληροφόρηση ξέρουμε ότι το να μπορεί κανείς να ελέγχει την πληροφορίες είναι κάτι το θεμελιακό είναι ο ακρογωνίας λίθος των αγορών μας και των οικονομιών μας του 21ου αιώνα. Αυτή λοιπόν, αυτός ο έλεγχος της πληροφόρησης, η προστασία της πληροφόρησης ε, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Η προστασία αυτής της πληροφόρησης, επαναλαμβάνω, των εγγύσεων των νομικών σε θέματα ε, που ανάφερα θα πρέπει να εξισορροπηθεί και με άλλα συμφέροντα και με άλλες αρχές ε, και αυτή την συζήτηση θέλουμε να ανοίξουμε και ανοίγουμε σήμερα για να μην ε, υποτιμούμε παράλληλα το, τα όλα τα λεπτά θέματα τα οποία τίθενται με αυτήν την έναρξη της συζήτησης για το σχέδιο οδηγίας τα θέματα της ε, ελευθερίας των συμφερόντων την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των επιχειρήσεων, ε, τον, του αντιφατικού χαρακτήρα του δικαίου σε ορισμένους τομείς. Όλα αυτά τα στοιχεία ε, μας οδηγούν σε μια αντιπαράθεση και σύγκριση τους ούτως ώστε να μπορέσουμε να μετακινήσουμε ορισμένες ισορροπίες. Και τελικά θέλουμε να οικοδομήσουμε μια τελική ισορροπία και να δούμε πώς θα τροπολοποιήσουμε το θέμα αυτό το πώς θα τροπολογήσουμε την οδηγία που έχουμε μπροστά μας, ούτω ώστε να διατηρήσουμε αυτή την, το πνεύμα εξισορρόπησης των διαφορετικών διακυβευμάτων και των διαφόρων ε, στόχων. Ο στόχος του κειμένου αυτού είναι να προσφέρει προστασία και εγγύηση για τις ε, εναντίον των παράνομων πρακτικών στον ανταγωνισμό και θέλουμε να ρυθμίσουμε ε, το, τις διάφορες ρυθμίσεις των σχέσεων των εταίρων ε, δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε τεράστιο βάθος αλλά γιατί είναι θέμα κρατών μελών από ένα σημείο και πέρα θέλουμε όμως να διατηρήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε θέματα τα οποία σαφώς ανήκουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα που δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες ε, της Ένωσης. Αυτή είναι η πρόταση. Η πρόταση θέλει να φτιάξει ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο. Ορισμένες διευκρινήσεις ε, τώρα για τους συναδέλφους που θα θελήσουν να λάβουν το λόγο στη συνέχεια. Υπάρχει μια ιδέα κύρια ε, την οποία αναφέρω για, να το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Μιλάμε για μια οδηγία η οποία ασχολείται με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων υποθέσεων. Δεν είναι αυτό αυτή η προσωνυμία του, του θέματος αλλά εν πάση περιπτώσει ε, η έννοια του μυστικού η ίδια μπορούμε να πούμε ότι θέτει προβλήματα ε, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα σε σχέση με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα και δημιουργούνται αντιδράσεις καμιά φορά έντονες, ε, συναισθηματικές θα λέγαμε. Ε, πρέπει να δούμε το κείμενο καθαρά, ξεκαθαρισμένα για να δούμε τι εννοούμε με τον μυστικό χαρακτήρα, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών υποθέσεων. Υπάρχουν διάφορες συμφωνίες πάνω σε ε, υπάρχουν σε ορισμένες χώρες εμπορικές συμφωνίες ε, και ο ορισμός δεν θέτει ένα πρόβλημα σε νομικό επίπεδο κατά την άποψή μου παρόλο που υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία ε, μπορούν να δημιουργήσουν κάποια θέματα στην αιτιολογική σκέψη ή σε ορισμένα άρθρα. Ειδικά το θέμα της εμπορικής αξίας για παράδειγμα θα έπρεπε ε, καλύτερα το, να διευκρινιστεί το τι είναι εμπορική αξία. Μετά υπάρχει το θέμα του αντικειμένου των άρθρων 3 και 4, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι εμπιστευτικές ε, υποθέσεις που πρέπει να προστατεύονται στον εμπορικό τομέα. Το, τα σημεία 3 και 4 μιλάει για νόμιμες ε, ε, οι ιδιοκτησίες και για παράνομες βέβαια εδώ δεν υπάρχουν ε, απριόρι σε σχέση με αυτούς τους ορισμούς αλλά βεβαίως μπορούμε να εισάγουμε κάποιες διευκρινήσεις και να ε, φτιάξουμε μια καλύτερη ισορροπία για τα θέματα αυτά. Η προστασία είναι σημαντική του μυστικού, το, το εμπορικό μυστικό δεν, ε, παν, δεν, έχει, δεν θα μείνει πάγια πάντα μυστικό, έτσι δεν είναι. Οπότε υπάρχουν ορισμένα μέσα τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ε, και να εφεύρουμε ορισμένα πράγματα. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να ε, προσδιορίσουμε περαιτέρω τη φύση των εργασιών μας. Χαίρομαι πολύ εκ των προτέρων για τις, τα σχόλια των συναδέλφων και πολύ καλή συνεργασία είχαμε τους συνεισηγητές. Κύριε Πρόεδρε, για το χρονοδιάγραμμα θα σας ζητούσα να μου, μας πείτε κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, και μετά θα έχουμε μια επόμενη συνεδρίαση γύρω στις 11 Νοεμβρίου και μετά ε, έχουμε την επιθυμία να προχωρήσουμε σχετικά γρήγορα, να μην χάσουμε χρόνο, αλλά Βεβαίως επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός παρεβενόντων και συμμετεχόντων που θέλουν να εκφραστούν ε, κοντά στις πολιτικές ομάδες και να μιλήσουν με τους εισηγητές, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας για τη διαβούλευση και για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις διάφορες απόψεις των εταίρων που ε, ε, θέλουν να συμβάλλουν στη συζήτηση και θέλουν να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. Ακούσαμε ήδη πολλούς, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί εταίροι τους οποίους δεν τους ακούσαμε και θέλουν να ε, έρθουν κοντά στα μέλη της Επιτροπής μας που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Το επόμενο σημείο, θα, η επόμενη συνάντηση θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο. Θα γίνει μια δημοσίευση του ώστε να μπορέσει να μεταφραστεί το κείμενο και θα, θα μεταφραστεί και στην ε, γλώσσα μου, ελπίζω τη μητρική πριν από τα Χριστούγεννα πριν από τις διακοπές. Μετά λοιπόν θα έχουμε την παρουσίαση της έκθεσης γύρω στη 19 η και 20 Ιανουαρίου για τροπολογίες. Μετά φαντάζομαι ότι θα πάμε στο Φεβρουάριο για τις τροπολογίες. Είναι βέβαια ένα σύντονο ε, χρονοδιάγραμμα αλλά δεν είναι υπερβολικά γρήγορο. Ε, ε, θα υπάρξουν λοιπόν οι τροπολογίες που θα συζητηθούν γύρω στις 23 με 24 Φεβρουαρίου. Εάν κρατηρήσουμε αυτές τις προθεσμίες θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε, να περάσει δηλαδή τον Μάρτιο η εισήγηση. Αυτά ήθελα να πω και σε αυτή τη φάση το χρονοδιάγραμμα αυτό θα μας επιτρέψει να περάσουμε στις επόμενες φάσεις. Έχουμε την θέση του Συμβουλίου που δούλεψε σύντομα και γρήγορα μέσα σε ένα θετικό εμψυχωτικό κλίμα και το σημειώνουμε αυτό. Επίσης έχουμε την δυνατότητα να καταρτήσουμε ένα κλίμα που θα μας δώσει την τη δυνατή συνένεση μέσα από το διάλογο. Σας ευχαριστώ συνάδελφε που πολύ αναλυτικά μας παρουσιάσατε όλες τις σημαντικές πλευρές αυτής της υπόθεσης η οποία είναι σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχ, προτείνω λοιπόν την εξή μέθοδο. Θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για να μας δώσουν τις δικές τους απόψεις. Μιας και έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση σας ακριβώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι τμήματάρχης για την καταπολέμηση των παραβάσεων στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς. Από ό,τι γνωρίζω η Γενική Διεύθυνση αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων και θα αποτελέσουμε τμήμα της νέας Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς. Το βασικό είναι να μείνετε στη δουλειά σας και να παραμείνει και η, διεύθυνσή σας, λέει ο κ. Καβαντά. Λοιπόν, μιας και η παρουσίαση είναι αγγλικά, θα παρουσιάσω και εγώ την δική μου παρουσίαση στα αγγλικά. Θα κάνω και εγώ τη δική μου παρουσίαση στα αγγλικά. Όπως η κυρία Λογρύπη ήδη εξήγησε, τα εμπορικά απόρριτα στοιχεία είναι ε, βασικά και για τις μικρές και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και θα επιμείνω στο θέμα των ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ε, σε υστερότερη φάση. Χρησιμοποιούν το θέμα της εμπιστευτικότητας σαν ένα μέσο διαχειριστικό για την ανάπτυξή τους. Βασίζονται σαν αυτά μυστικά για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους και εκτιμούν τα εμπορικά αυτά μυστικά ακόμα περισσότερο και από τις ίδιες τις ευρεσιτεχνίες. Όπως είπε η κυρία Γκρίπη υπάρχει μια επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία. Τα εμπορικά μυστικά από τη μία και τις ευρεσιτεχνίες από την άλλη. Κάθε δικαίωμα έτσι κι αλλιώς συγγενικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ξεκινά σαν ένα εμπορικό μυστικό πριν από οτιδήποτε άλλο. Το βασικό για μας είναι να παίξουν αυτά τα εμπορικά μυστικά ένα σημαντικό ρόλο στη σώρευση γνώσεων ανάμεσα σε εταίρους, σε επιχειρήσεις και στο εσωτερικό της ε, αγοράς μας. Είναι σημαντικός ο ρόλος λοιπόν αυτών των παραγόντων στον τομέα της ε, ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Ο συνδυασμός και η συνδυασμένη έρευνα είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ιδιαίτερα σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον εμπορικό και είναι βασικό για να αυξηθεί η έρευνα στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Αυτά είναι τα θετικά. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη έκθεση σε καταχρηστική μεταχείριση αυτών των μυστικών. Κάναμε δύο έρευνες η μία αφορά την ετήσια έκθεση για τη βιομηχανία στο εσωτερικό της ετήσιας αυτής έκθεσης, ε, δηλαδή ένας κατάλογος ε, βιομηχανιών και επιχειρήσεων ε, από το σύνολο του φάσματος της παραγωγικής δραστηριότητας και εταιρείε οι οποίες έχουν τύχει στο παρελθόν ε, προβληματικών χρήσεων στον τομέα των μεθόδων που δημιούργησε προβλήματα στις επιχειρήσεις αυτές. Η κλοπή πληροφοριών από το 2008 μέχρι το 2013 αφορούσε το 18% των επιχειρήσεων και είχε φτάσει το 2013 γύρω στο 25%. Βλέπετε δηλαδή ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που θίγεται από, αυτό το φαινόμενο αυξάνεται. Τώρα, για την εσωτερική αγορά. Όπως παρατήρησε ήδη η κυρία Λεγκρίπ, έχουμε την συμφωνία η οποία απαιτεί από τους συμμετέχοντες να προστατεύουν αυτά τα εμπορικά μυστικά. Ελπίζω η διαφάνεια αυτή να είναι αναγνώσιμη από τα μέλη <clears throat> κάτω αριστερά, βλέπουμε ότι υπάρχουν ένα patchwork, διαφορετικά επίπεδα προστασίας στις χώρες μέλη. Βλέπετε ότι κάθε χώρα μέλη έχει κάποια από τα στοιχεία της προστασίας τα οποία είναι προαπαιτούμενα, από την άλλη όμως υπάρχουν και κάποια άλλα, τα οποία ελείπουν. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι κάποιες χώρες δεν έχουν καν νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι με κανένα τρόπο δεν τα προστατεύουν αλλά αυτό το κάνουν με βάση το απλό αστικό δίκαιο και την αστική νομολογία στη συγκεκριμένη χώρα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει προστασία απέναντι σε τέτοιου είδους καταχρήσεις, αλλά μόνο σε σχέση με ανταγωνιστές και όχι σε σχέση με άλλους τρίτους. Και δεν υπάρχουν επίσης και δυνατότητες αποζημίωσης σε πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι πάντα δυνατό λοιπόν σε ένα κράτος μέλος και στα πλαίσια των διαδικασιών των εθνικών να διατηρήσει κανείς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Το πρόβλημα λοιπόν όπως το βλέπουμε εμείς είναι ότι η εσωτερική αγορά είναι πράγματι ε, σε δύσκολη θέση λόγω αυτής της πολυδιάσπασης της μορφής προστασίας και της έλλειψης διαφάνειας. Όπως είπα νόμοι υπάρχουν το θέμα είναι όμως ότι ποικίλει η κατάσταση ανάλογα με το που βρίσκεσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάρα πολύ δύσκολο συνολικά να κατανοήσει κανείς ποιες είναι οι νομικές μορφές προστασίας των συμφωνιών που κάνει μια επιχείρηση. Το 40% των επιχειρήσεων με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή είπαν ότι δεν θα μοιράζονται τέτοιες πληροφορίες διαμεθοριακά δεν θα αναζητήσουν δηλαδή τους ιδανικούς επιχειρηματικούς εταίρους σε άλλες χώρες, λόγω των φόβων που έχουν. Και ε, άνω του 50% των επιχειρήσεων είπαν ότι αυτές οι δραστηριότητες, αυτό το φαινόμενο υπονομεύει τις ε, διεθνείς εμπορικές τους συναλλαγές. Θα σας τα δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία με πιο αναλυτικό τρόπο. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε τώρα. Νομίζω ότι στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καταχρηστική μεταχείριση των εμπορικών μυστικών, των επιχειρηματικών μυστικών και να βελτιώσουμε τις συνθήκες για μια σωστή εκμετάλλευση της καινοτομίας στο εσωτερικό της Ένωσης. Επίσης, προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών επιχειρήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες είναι ε, ο πυρήνας της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, είτε είναι μια μικρή startup, είτε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εμείς δεν προτείνουμε εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπαρκές. Η Συμφωνία TRIPS ε, είναι σε ισχύ εδώ και 20 περίπου χρόνια και αν ενθυμίστε τη διαφάνεια που σας ένδειξα υπάρχει μια πολυδιάσπαση στα κράτη-μέλη. Και στο τομέα της ε, πολιτικής προστασίας ε, και σε σχέση με το αντίστοιχο άρθρο. Έρχομαι τώρα στην οδηγία αυτή που όπως είπε η κυρία Λεγκρίπ έχουμε έναν ορισμό όσον αφορά την συνεκτικότητα και συμβατότητα με τις διατάξεις. Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε τον ορισμό του εμπορικού απορρίτου και που πρέπει να αφορά και τον ορισμό του τι είναι παράνομο. Και θα δείτε λοιπόν στο τετραγωνάκι το κόκκινο στη δεξιά πλευρά της οθόνης, δεν θα επισέτω περισσότερο, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου όσον αφορά τα θέματα της ε, χρήσης αποκάλυψης στοιχείων από τρίτους ε, ενώ θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για απόρριτα ή για ηχέμηθα στοιχεία. Είναι σημαντικό <clears throat> σε σχέση με κράτη-μέλη η διασφάλιση αυτής της προστασίας ε, και θέματα παραβίασης ή παράβασης ώστε να μπορεί να αναλυθεί δράση σε σχέση με όσους παραβιάζουν ή παραβαίνουν αυτές τις αρχές. Επίσης ε, έρχομαι σε ένα σημείο που προηγούμενα αναφέρθηκε και αυτό που κάνουμε είναι με αυτή την πρόταση, το άρθρο 4, το πρώτο παράδειγμα για την ισορροπία που θέλουμε να επιτύχουμε, καθορίζουμε με σαφήνεια όσον αφορά το τι μπορεί να είναι το νόμιμο πλαίσιο. Δηλαδή λέμε ότι δεν ασχολούμεθα με αποκλειστικά θέματα ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και θα πρέπει εδώ να λαμβάνετε υπόψη το θέμα της ε, νομικής ε, υπόστασης αυτών των θεμάτων για την αποσαφήνιση τους. Και σε σχέση με το άρθρο 4.2 εξαιρέσεις ε, όσον αφορά άλλα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης για παράδειγμα. Επιτρέπουμε και θέλουμε να διευκολύνουμε την ε, αποκάλυψη πληροφοριών από πληροφοριοδότες ε, whistleblowers ε, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα στοιχεία και αυτά τα στοιχεία που μια επιχείρηση δεν θα ήθελε να αποκαλύπτονται πρέπει εδώ να λαμβάνονται υπόψη. Έρχομαι τώρα σε θέματα επανόρθωσης ή αποζημίωσης. Αυτά είναι συγκεκριμένα θα έλεγα. Εδώ πρόκειται για συγκεκριμένους τύπους, ε, για παραβίαση ε, συγκεκριμένων θεμάτων όπου θα έπρεπε να λαμβάνονται τέτοια μέτρα επανόρθωσης. Και έχουμε και εναλλακτικά μέτρα αντιστάθμισης ή επανόρθωσης και πάλι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αναλογικότητα στην εφαρμογή όλων αυτών. Να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά τη ζημία που θα έχει προκληθεί με την αποζημίωση που θα καταβάλλεται. Ένας άλλος τομέας διασφαλίσεων που έχει και αυτό στη σημασία του, όπως προανέφερα, είναι απόλυτα θεμελιώδους σημασία σε αυτόν τον τομέα, κάτι το οποίο απορρέει με απόλυτη σαφήνεια σε σχέση με τη διαβούλευση που είχαμε και κάναμε με επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους σημασία σε σχέση με θέματα νομολογίας θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε σχέση με τέτοια πληροφοριακά στοιχεία. Αλλά αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων ορισμών και περιπτώσεων. Συχνά τέτοιου είδους εμπορικά απόρριτα δεν, ε, είναι, ε, δεν αποκαλύπτονται και θα διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν ρήτρες ε, διασφάλισης, δικλίδες ασφαλείας για την κάλυψη και διασφάλιση αυτών των στοιχείων όταν θα υπάρχει ένα τέτοιο επίμαχο θέμα. Είναι ένα θέμα ρήτρα διασφάλισης που έχει την σπουδαιότητά του. Επίσης έχουμε και ένα όριο περίοδου παραγραφής καθορίζουμε ότι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο χρόνια. Δύο χρόνια μετά την ε, παραβίαση διατάξεων ή την αποκάλυψη παραβίασης τέτοιων διατάξεων. Και πάλι ο λόγος γι' αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι μετά από δύο χρόνια <clears throat> όταν θα έχει γνωστοποιηθεί ότι υπήρξε παραβίαση, αν το εμπλεκόμενο μέρος δεν έχει αναλάβει δράση, ε, τότε λοιπόν ε, δεν θα μπορεί μετά από δύο χρόνια να αναλυθεί δράση για την ε, παρακόλληση περαιτέρω αποκαλύψεων. Και υπό τους όρους εν τέλει και θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Είχαμε επίσης και συμπληρωματικές διατάξεις εποπτείας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της ε, οδηγίας. Πρόγραμμα, για παράδειγμα, για την ε, διασφάλιση της ε, ένταξης αυτών των διατάξεων στην καλύτερη νομοθετική πρακτική. Και τέλος, και επιτρέψτε μου εν συντομία να τα αναφέρω πρόεδρε, πρόκειται για μια επισκόπηση της ωφέλειας που θεωρούμε ότι δημιουργείται εδώ, του ωφέλους που δημιουργείται και από πλευράς της ε, κυρία Λεγκρίπ ε, τονίστηκε η σπουδαιότητα. 77% των επιχειρήσεων είναι υπέρ της ε, καλύτερης προστασίας των εμπορικών απορρίτων. Και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που σε σχέση με διαδικαστικά θέματα θεωρούν ότι θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας. Και επίσης 63% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι αυτό θα πρόσφερε περισσότερες καλύτερες ευκαιρίες ε, για θέματα ε, πρόθεσης νοτομίας και 49% είναι υπέρ της ε, κοινή εκμετάλλευσης έβρεση τεχνιών και ολοκληρώνω και ελπίζω ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνεννοηθούμε. Είναι η κοινή δημόσια διαβούλευση αυτή και τα αποτελέσματα αυτής θα δείτε ότι εφιστώ την προσοχή σε δύο σημεία. Πρώτο, αν δείτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι συμβαίνει με αυτές. 73% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απάντησαν είπαν ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με ρυθμιστικά πλαίσια και κανονισμό, κανονισμούς. Είναι αυτό υψηλού επίπεδου προστασία. Έχουν, ανησυχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις υπερβολικές ε, ρυθμιστικές διατάξεις ε, και το εύρος τους. Και αυτό δείχνει ότι είναι, έχει τη σημασία του αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης αποκαλύπτει το γεγονός και θα δείτε σε αντιδιαστολή με αυτό μόνο 19% από όσους απάντησαν σε σχέση με αυτή την πρόταση εξέφρασαν την ίδια γνώμη. Και αυτό τι δείχνει. Δείχνει με σαφήνεια την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση για το τι τεκταίνεται από πλευρά μα. Και γι' αυτό καλωσορίζουμε την ευκαιρία το Κοινοβούλιο να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί και να κινητοποιηθεί. Και πάλι όμως θα ήθελα να τονίσω αυτά τα στοιχεία σε εσά. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό για την ε, α, ανάλυση επιχειρήσεων, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα δείτε ότι είναι υπέρ της νομικής ρύθμισης και μόνο 17% κατά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπερζοβά. Ευχαριστώ και για τις ενδιαφέρουσες διευκρινήσεις τις οποίες κάνατε. Δύο επιπλέον πληροφορίες και μία ερώτηση. Η ερώτηση. Τι εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, δυνατότητα ύπαρξης ε, ενός κοινοτικού κανονισμού και όχι άλλων μορφών ρυθμίσεων. Η δεύτερη ερώτηση είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε αργότερα, δηλαδή θα του ζητήσουμε από τους συναδέλφους να πάρουν το λόγο γύρω από αυτό, αλλά μιας και δεν είμαι ε, παραευκαιριακός προεδρεύων, θα ήθελα και σαν συντονιστής να εκφράσω και εγώ την άποψή μου, ελπίζω αυτό να μην σας ενοχλήσει. Τρίτον, θα μου πείτε αν συμφωνείτε και θα ξεκινήσω από αυτό, να <clears throat> κάποιοι από εμά, μεταξύ των οποίων και η ίδια η κυρία Λεγκρίπ, να οργανώσουμε μία ακρόαση, γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Και όταν βλέπουμε τα ποσοστά στα οποία αναφερθήκατε των θυγωμένων επιχειρήσεων, Διαπιστώνουμε ότι εδώ υπάρχει προσδοκία κοινοτική. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, γιατί να μην υπάρξει μια ενιοποίηση ευρωπαϊκή. Σας ελείπει η νομική βάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σαφής. Προσπαθούμε να αναβωνήσουμε αυτή τη φάση, το κάνουμε, κάποιες διαδικασίες αστικού δικαίου. Και πιστεύουμε και αυτό ισχύει για τα αποκλειστικά δικαιώματα, υπάρχει μια οδηγία η οποία έχει προχωρήσει σε εναρμόνιση και πιστεύουμε ότι ένας κανονισμός θα ξεπεράσει το τι είναι απαραίτητο. Ε, γιατί τελικά πάντα τα δικαστήρια θα είναι αυτά κατά περίπτωση να κάνουν τις εκτιμήσεις τους ε, γύρω από τα θέματα της αναλογικότητας κτλ. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι υπερβολικό στην παρούσα φάση ένας κανονισμός, γιατί ε, στην ουσία θα δεσμεύαμε, θα παγώναμε με αρνητικό τρόπο, ε, όπως λέει ο νομοθέτης, θα περιορίζαμε αν θέλετε ε, τις δυνατότητες που έχουν οι δικαστές, οι νομικές, οι κριτές. Κυρία Ρέγνα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση από την Επιτροπή και από πλευράς της κυρίας Λεγκρίπ για την παρουσίασή της για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Τον κύριο Κοφεράτη ε, εκπρόσωπο <clears throat> και οδησηγητή για τους σοσιαλδημοκράτες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε συνέχεια στο θέμα των εμπορικών ε, ε, απορρίτων γιατί αυτά τα θέματα θα είναι κύριος στόχος του 21ου αιώνα. Πρέπει να προστατέψουμε ιδιαίτερα τα θέματα τα οποία πρέπει να προστατευθούν. Και κατά τούτο είναι σαφές πλέον ότι όταν έχουμε ενώπιον μας καταστάσεις νομικές στα κράτη-μέλη που αφορούν αυτά τα θέματα, όταν υπάρχουν νομικές αβεβαιότητες ή ανασφάλεια, λόγω διαφορετικών καθεστώτων που ισχύουν από χώρα σε χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να το λάβουμε υπόψη και πρέπει να καλωσορίσουμε το γεγονός ότι υποβάλλει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά ώστε να υπάρξει πρόσθετη αξία για την Ευρώπη. Ένα πράγμα πρέπει να αποσαφινιστεί θεωρούμε εμείς συγκεκριμένα και εξειδικευμένα όταν κάνουμε λόγο για το νομοθετικό έργο και όταν κάνουμε λόγο για πνευματικά δικαιώματα, πραγματικά οι δικαιούχοι να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους νομοθετικές προτάσεις και διατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό όταν συζητούμε θέματα εμπορικού απορρίτου να το λάβουμε αυτό υπόψη αλλά ακόμα και για μια δεύτερη κατηγορία δικαιώματα. Όταν έχουμε εδώ λοιπόν λόγο για διαφορετικά θέματα και τα θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις ε, επιχειρήσεις μας ε, και που κάποιοι μπορούν ίσως παράνομα να προμηθεύονται και αυτό μπορεί να αποβαίνει εις βάρος των επιχειρήσεων. Όλα εξαρτώνται από το πώς θα προσεγγίσουμε σφαιρικά αυτό το θέμα για να προστατεύονται αυτά, αυτές οι πληροφορίες και να δραστηριοποιηθούμε ώστε οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη να μπορούν πραγματικά να προστατεύονται στο πλαίσιο λειτουργίας τους για να στεφθούν με επιτυχία οι δράσεις τους. Εμείς θεωρούμε ότι τα εξής πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εξετάζουμε με ιδιαίτερη, με ιδιαίτερη προσοχή τους ορισμούς. Οι ορισμοί λοιπόν θα πρέπει να επικεντρώνονται με ιδιαίτερη σαφήνεια σε ένα σαφές πλαίσιο ώστε να καταπολεμούνται οι περιπτώσεις ε, ε, ανομίας ή παρανομίας και της παράνομης απόκτησης ε, πληροφοριών. Και μια δεύτερη συνιστόσα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ο ρόλος των εργαζομένων στις επιχειρήσεις γιατί κατά το μάλλον ήταν είναι ακριβώς οι εργαζόμενοι, οι απασχολούμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις ως φορείς αυτών των στοιχείων, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούν ίσως να μεταφέρουν ή να διοχετεύουν τέτοιου είδους ε, στοιχεία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν εξετάζουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Να λάβουμε υπόψη τα εξής στοιχεία. Έχουμε χώρες όπως την Γερμανία ή την Αυστρία όπου εκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια οι εργαζόμενοι και έχουν και πάλι στη διάθεσή τους πολλά πληροφοριακά στοιχεία, διότι μέσω της δραστηριότητάς τους δουλειά τους είναι επίσης να διαχέονται αυτές οι πληροφορίες και να διοχετεύονται και προς τους άλλους εργαζόμενους. Έχουμε ένα πεδίο εντάσεων λοιπόν εδώ όπου θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού ξεκινά, ποια είναι η γένεση ενός ε, εμπορικού απορρίτου και πώς αυτό εξελίσσεται ώστε να μπορεί να προστατεύεται. Και μέσα στο πλαίσιο της ε, λύσης, της πρότασης αυτής ε, γενικότερα να κάνουμε μια ακρόαση ώστε να λάβουμε υπόψη τα πιο διαφορετικά στοιχεία τα οποία ενέχονται. Αυτά σε σχέση με αυτές τις δύο πρώτες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. La Ευχαριστώ. Το λόγο Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ αυτό το θέμα τεράστια σημασίας Πρόεδρε. Και αυτή η σπουδαιότητα ακριβώς βρίσκεται και στην προηγούμενη παρέμβαση από πλευρά συναδέλφου και της εισηγήτριας ε, για αυτό το θέμα. Η προστασία του εμπορικού απορρίτου έχει μια οικονομική αξία που πρέπει να, προασ... να την υπερασπιστούμε και να την προστατευτούμε όσον αφορά τις νομικές διατάξεις και τα νομικά πλαίσια των κρατών μελών. Μέσα από ένα εμβριώδες ε, μόρφωμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αποκρισταλώσει τον πολιτικό της στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση αν είναι σε θέση να κάνει ένα βήμα για να διασφαλίσει ότι θα μπορούν μέσα από αυτό το πλαίσιο νομικής διασφάλισης ε, να προστατεύουν οι νομικές πτυχές ε, από πλευράς δικαιώματος Τώρα, για το θέμα της προστασίας της ίδιας του ίδιου του εμπορικού απορρίτου εμπορικών επιχειρήσεων και εταιριών, εδώ έχουμε και το θέμα της, του απόρριτου, του επαγγελματικού απορρίτου και του βιομηχανικού επιχειρησιακού απορρίτου. Η προστασία λοιπόν αυτού του αγαθού, αυτής της αξίας, έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία στο σημερινό κόσμο και θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να δούμε τι θα μπορεί να γίνει αν υπάρξει ακριβώς ε, το πλαίσιο ώστε να κυρώνονται, να υπάρχουν, να, να κολλάζονται άμεσα, να τιμωρούνται οι πράξεις ε, εκείνες που παραβιάζουν και παραβαίνουν αυτές τις νομικές διατάξεις προστασίας αυτών των αγαθών. Η παραβίαση ενός ε, εμπορικού απορρίτου και η απλή παραβίαση κανόνων του ανταγωνισμού ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, ή το λάδωμα ε, κάποιων που ε, μπορούν χρηματικά ε, με κάποια χρηματικά δώρα τα οποία παίρνουν να αποκαλύψουν κάποια στοιχεία όλα αυτά δίνουν λοιπόν αυτό το πλαίσιο η ε, κοινοί γνώμη, οι ε, πολίτες μας λοιπόν πρέπει να δούμε σε σχέση με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις να δούμε ότι σε σχέση με την διαβούλευση είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι στάσεις και οι θέσεις αυτές. Και γιατί, διότι γενικά συνδέεται η προστασία ακριβώς αυτών των θεμάτων με την προστασία την υπερβολική ή η καταχρηστική προστασία που καμιά φορά μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης θέσης μιας επιχείρησης στην αγορά και που για παράδειγμα για τα ιατρικά προϊόντα, για τα φάρμακα και για την απόκτηση μεγαλύτερου κέρδους από μια επιχείρηση ε, μέσω της διοχέτευσης των προϊόντων τους. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια να συγκλίνουν ε, τα ε, συμφέροντα των πολιτών και σε σχέση και με το πώς θεωρούν οι πολίτες αυτά τα θέματα. Είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να δράσει, να δώσει, να κάνει θετικά βήματα ώστε να παγιώσει, να ολοκληρώσει αυτό το εγχείρημα από από νομικής πλευράς. Είναι ανάγκη να υπάρξει ένας ε, νομικός εναρμονισμός ε, από πλευράς των κρατών μελών. Στις διάφορες αυτές νομικές διατάξεις ε, και φάσεις για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται αυτά τα θέματα από κράτος σε κράτος, ώστε να μπορέσουν αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πιο γενικό εναρμονισμένο πλαίσιο να λειτουργήσουν. Αυτό είναι το αναγκαίο που πρέπει να γίνει. Να κάνουμε βήματα για να προχωρήσουμε στην παγίωση μιας νομικής τάξης πραγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Οι σα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό αγαπητέ συνάδελφοι. Άλλε παρεμβάσεις, παρακαλώ. Πράγματι είναι χρήσιμη αυτή η νομοθετική ρύθμιση η προτινόμενη είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα της καινοτομίας. Είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει. Ε, ξέρω ότι πολλοί ασχολούνται με το θέμα αυτό και ίσως σε 20 χρόνια να βρεθεί μια κάποια λύση. Θα ζητήσω από την Επιτροπή και τον εισηγητή να εξετάσει το άρθρο 3 του συγκεκριμένου κειμένου στο σημείο 2 του άρθρου 3 η απόκτηση ενός επιχειρηματικού μυστικού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου ή σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις στην προστασία του επιχειρηματικού απορρίτου. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να οριστούν κάπως καλύτερα. Θα πρέπει να ορίσουμε με σωστότερο τρόπο το ποιος είναι υπεύθυνο όταν αποκτά ένα τέτοιο επιχειρηματικό μυστικό. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε την Επιτροπή και τον εισηγητή που έκανε την εισαγωγή σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Να επανέλθω στη σχέση σε σχέση με, τα εμπορικό, με το εμπορικό απόρριτο και τις, ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι πολύ σημαντικό να μην, υπονομεύονται, να μην υπονομεύονται οι στόχοι της ε, δημόσιας ε, πολιτικής. Όταν υποβάλλει κάποιος μια αίτηση για ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το κράτος δίνει κίνητρα ίσως ε, για να υπάρξει αποκάλυψη κάποιων στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν σε καινοτομία από άλλες επιχειρήσεις και σε αντάλλαγμα επιχειρήσεις ε, παίρνουν ένα είδους μονοπόλιο στην εκμετάλλευση κάποιων στοιχείων τα ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και της, ε, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε έναν ανταγωνισμό που μπορεί να δημιουργείται. Θα πρέπει να προχωρούμε με την με, με, με ένα σήμα εμπορικό ή με ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χωρίς όμως να υπάρχει υπονόμευση του συστήματος που λειτουργεί στην Ευρώπη. Να διασφαλίσουμε δηλαδή να υπάρχουν κίνητρα για εταιρείες, για εταιρείες ώστε να μπορούν να αποκαλύψουν κάποια στοιχεία ώστε να αποτελέσουν αυτά κίνητρα να δραστηριοποιηθούν άλλες εταιρείες. Κάτι άλλο που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διατυπώσεις στο άρθρο 4 σε σχέση με τις ε, ε, εξαιρέσεις ε, και για την νόμιμη χρήση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης. Αυτό το νόμιμος legitimate δημιουργεί ένα υψηλό φραγμό για την ελευθερία πληροφόρησης και ενημέρωσης για ένα αντεπιχείρημα για παράδειγμα για την διασφάλιση του εμπορικού απορρίτου στο γερμανικό πλαίσιο χρησιμοποιείται το, ο όρος νόμιμος ως ε, ορισμός. Μόνο όταν υπάρχει ένα νόμιμο ε, κίνητρο ή ε, ένα, ένας νόμιμος λόγος μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα. Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα μη αδειοδοτημένο χημικό, μια μη αδειοδοτημένη χημική ουσία, τότε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παραβίαση εμπορικού απορρίτου. Στον ορισμό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές ε, για τα νόμιμα θεμητά συμφέροντα από πλευράς ε, εμπορικών απορρίτων, από πλευράς των επιχειρήσεων. Αντί να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει νόμιμο συμφέρον για οποιονδήποτε που αποκαλύπτει ένα τέτοιο εμπορικό απόρριτο χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της ελευθερίας της έκφρασης. Κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε και αυτό λίγο περισσότερο να αποσαφινιστεί είναι το ότι δεν κάνουμε λόγο για ένα αποκλειστικό δικαίωμα ιδιοκτησίας και πραγματικά πολλά κράτη-μέλη υπό αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζουν το εμπορικό απόρριτο μέσα στο πλαίσιο του, της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό για παράδειγμα, ή για την κατάχρηση ε, τέτοιου είδους ε, ε, δικαιωμάτων. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν <clears throat> ότι σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις τα θέματα εμπορικού απορρίτου πρέπει να συζητούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα θέλαμε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρότασή της ως έχει αποτελεί τη βάση για τις διαπραγματεύσεις, ε, τη διαπραγματευτική βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη Συμφωνία Εμπορικών Σχέσεων και Επενδύσεων με τις ΗΠΑ, TTIP και να μας πείτε επίσης σε σχέση με το πλαίσιο αυτό είναι ένα είδους ε, ε, εμπορικής συμφωνίας ή εμπορικού απορρίτου. Είναι διαφορετικό από τα δικαιώματα IPR ή για τα θέματα ε, συμβόλων, εμπορικών συμβόλων, trademarks. Μήπως αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια διαφορά σε σχέση με την πρόταση που υποβάλλεται Εν τέλει θα ήθελα να με ενημερώσετε, να καλωσορίσω την πρόταση από πλευράς εισηγητού να διεξαχθεί μια ακρόαση για αυτό το θέμα και να συμπεριληφθεί και το θεμελιώδες δικαίωμα για αυτό το χαρτοφυλάκιο να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την προστασία των εμπορικών ε, απορρίτων που δεν θα υπονομεύει όμως τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε σύντομα ε, σε αυτή την ερώτηση σας παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με δύο σημεία που έθιξε η κυρία Ρέντα το ένα η νόμιμη χρήση της ελευθερίας έκφρασης, κατανοώ την θέση της. Ε, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τη λογική της ελευθερίας της έκφρασης ε, στην νομολογία αυτής της χάρτας. Πρέπει να την κρατήσουμε όσο πιο ευρία γίνεται. Αυτό επιθυμούμε. Το δεύτερο ε, ερώτημα σε σχέση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρούσα στιγμή που βασίζεται σε αυτή την πρόταση, δεν διαπραγματευόμαστε αυτή την πρόταση, τώρα έχει εγκριθεί, είναι σαφές αυτό ε, και η θέση μας είναι ότι δεν είναι αποκλειστικό το δικαίωμα, ότι από την άλλη πλευρά ε, ίσως υπάρχει ένα διπλό σκέλος που καλύπτει ε, ε, τα θέματα όλα της ευρεσιτεχνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν έχει παρέμβει σε αυτό το σημείο και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. και εγώ ζητώ άδεια από τους συναδέλφους μου να εκφραστώ ως συντονιστής αγγε για να θίξω αυτά που υπόθηκαν σε, στις περισσότερες παρεμβάσεις και στην τελευταία μάλιστα να μην επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν για να μην χάσουμε χρόνο σε σχέση με την σημασία τη μεγάλη το, του να καταρτιστούν πρακτικές ε, ε, και να εναρμονιστεί όσο περισσότερο γίνεται το πεδίο αυτό στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Θα ήθελα να πω επίσης δύο πράγματα. Το κεντρικό σημείο που να ληφθεί υπόψη για μένα είναι η απουσία συγκατάθεσης ε, των χρηστών αυτής της υπόθεσης όπου γίνεται παράβαση γίνεται μια πρόσβαση, ε, μια κλοπή, μια πρόσβαση που δεν έχει πάρει άδεια, ε, μια κατάχρηση εμπιστοσύνης, μη σεβασμός μιας συμφωνίας ε, απορρίτου και με δύο λόγια αυτή η συμπεριφορά που έχει σχέση με την χρήση την εμπορική δεν είναι έντιμη. Πρέπει κάθε τέτοια συμφωνία να, είναι, να χαρακτηρίζεται από εντιμότητα. Έτσι χρειάζεται να υπάρχει άδεια για την παροχή υπηρεσιών, τη διάδοσή τους, τη μετάδοσή τους ε, και χωρίς να ε, γίνεται ανάμιξη ε, των διαδικασιών που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη, ε, παρόλο που σε μερικά κράτη-μέλη υπάρχουν παρόμοια σημεία. Στην ενία αγορά υπάρχουν νόμοι για την πνευματική ιδιοκτησία και πρέπει να υπάρξει ένα καθεστώς προστασίας τους. Είναι απόλυτα νομότυπο το να υπάρχει συμπλήρωμα σε αυτή τη νομοθεσία. Ενθαρρύνω βεβαίως όλες αυτές τις προσπάθειες και σε σύμφωνη γνώμη με την εισηγήτρια να και με την άδεια σας αγαπητοί συνάδελφοι γιατί εσείς θα εγκρίνετε σε τελική ανάλυση ή θα απορρίψετε να καταρτήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες σχετικά γρήγορα και πριν να κατατεθεί, ε, κατατεθούν οι τροπολογίες μιλήσατε για την 23η 24η είπατε για αρχές Φεβρουαρίου 27 ε, ε, Φεβρουαρίου είναι μια ημερομηνία που μου είναι πάρα πολύ προσφύλης αν το θυμάστε. Ε, εν πάση περιπτώσει είπαμε να κάνουμε μια δημόσια κρόαση πάνω σε αυτή την απόφαση που να έχει μεγάλο εύρος όσο πλατύτερο γίνεται για να μπορέσουμε να έχουμε μια κάλυψη όλων των σημαντικών θεμάτων το τι βλάβη υφίστανται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις μέσα στην Ήπειρό μας παρόλο που οι μεγάλες προστατεύονται καλύτερα με εσωτερική προστασία, με γραφεία δικηγόρων κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε κάτι το επικοδομητικό πάνω σε αυτό το θέμα που ενδιαφέρει τους πελάτες και οι σφιγμομετρήσεις που κάνατε το αποδεικνύουν. Ποιοι είναι λοιπόν, ποιος είναι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης πάνω σε αυτό το θέμα να σηκώσει το χέρι. Κατά. Σήκωσε κάποιος το χέρι, κάποιος είναι κουρασμένος. Είναι κανείς κατά, κανείς. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημειώστε παρακαλώ κύριε Μπρέτ ότι σύμφωνα με την κανονική διαδικασία θα ζητήσουμε να περάσει στη διάσκεψη των Προέδρων το θέμα αυτό με αίτημα ακρόασης. Τώρα τα επόμενα σημεία, ποια είναι τα επόμενα σημεία που έχουμε να διεκπαιρεώσουμε. Αγαπητοί φίλοι, θα δουλέψουμε και κλεισμένων των θυρών για το επόμενο σημείο. Παρακαλώ να διάστε την αίθουσα.